Okay, colleagues, if people can start to take their seats now. Καθίστε παρακαλώ, συνάδελφοι, λέει η Πρόεδρος, να αρχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είχαμε την πρώτη κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Οπότε αρχίζει η δική μας συνεδρίαση τώρα. Άρα ουσιαστικά είναι το δεύτερο σημείο της σημερινής διάταξης έγκριση Αλλαγές δεν έχουν ε, προταθεί. Α, όχι, όχι, υπάρχει. Υπάρχει ο κύριος Βέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Of Η πολιτική μας ομάδα θέλει να αναβληθεί η αυριανή ψηφορία όσον αφορά τη λύση του χρέους των ψωμένων χωρών. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση από του συναδέλφου που έχουν λάβει το θέμα. Και έτσι να έχουμε περισσότερο χρόνο ε, να το μελετήσουμε το θέμα. Ζητούμε πνεύμα επομένω συμβαστικό. Τι λέει ο εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας εξηγήσω πώς οργανώσα τη δουλειά για την υπόθεση αυτή. 31 πρώτου ήταν το όριο για τις ε, τροπολογίες, όλα από το ήταν στα πολωνικά, οπότε και δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Όμως, στο μεταξύ προσπάθησα να οργανώσω συνάντηση των σχεδόν εισηγητών στο Στρασβούργο. Και θα είχαμε με τη μέθοδο του ψιθυρισμού διερμηνία όσον αφορά τους Πολωνούς συναδέλφους, αλλά αυτό όμως τελικά δεν εγκρίθηκε και επομένως ξεφύγαμε από το timing της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε τι να κάνω ως ε, εισηγητής δεν μπορώ να τηρήσω αυτά τα οποία αποφασίσαμε άρα τι να πω στο ΕΛΚ σε σχέση με το αίτημα τους εδώ και κάποιες μέρες μου τα είπανε είναι θέμα εμείς της διαταξής μας δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που είπε ο κύριος Βέντα φιλικά του το λέω. Ο Μπόγκταν πάντοτε ήταν εντάξει με όλα και έναντι όλων των συναδελφών. Αν δεν ήταν ο Μπόγκταν που να το ζητούσε αυτό θα είχα πει όχι. Γιατί πάρα πολλά αναλυθεί κυκλοφόρησαν μέσω emails τις τελευταίες μέρες. Προσπαθώ να καλύψω όσα ζητάνε όλοι γύρω γύρω αλλά μέχρι ενός σημείου επομένω. να το συζητήσουμε έστω και αν χάνουμε έτσι λίγο χρόνο επομένως γιατί σε, πνεύμα συμφιλίωσης να τα πούμε α λέει πρόεδρος ωραία δεν βλέπω καμία ένσταση τι λέτε Βέντα Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για τις εξηγήσει τον εισηγητή. Να σας τα πω στα γερμανικά, οπότε Ίσως είναι πιο άμεση η συνεννόηση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ νομίζω σε ενημέρωσα ότι την πράσινη αυτή εβδομάδα, την τυρκόσα εβδομάδα, υπήρχε αποστολή για τη Σενεγάλη. Το θέμα της μετάφρασης, της διερμηνίας, ε, ξέρουμε ότι υπήρχαν δυσκολίες, αλλά βεβαίως τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Μέχρι τώρα δεν είχαμε άλλες δυνατότητες και όντως δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε κατευθείαν ε, πρόσωπο με πρόσωπο και εδώ στην Επιτροπή είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την επικοινωνία και να διατηρήσουμε και το διάλογο. Ευχαριστώ πολύ πάντως για αυτά που είπες. Αν συμφωνείτε συνάδελφοι, να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την επόμενη συνάντησή μας. Θα μας πει η γραμματεία πότε, το συντομότερο δυνατόν. Το Μάρτιο, μου λέει η Ντονατέλα, θα γίνει αυτό. Έχω καταλάβει ότι αυτοί που πήγαν στην Σενεγάλη ήταν εφιαλτικό το ταξίδι της επιστροφής. Χαίρομαι που είστε εδώ Και ξέρω ότι κάποιοι που έπρεπε να είχαν επιστρέψει σπίτι τους την Παρασκευή έφτασαν σήμερα το πρωί. Mm. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά η αποστολή σας και εγώ επέστρεψα από την Κεφρική και νομίζω ότι θα πρέπει να ανταλλάξουμε πληροφορίες και να μιλήσουμε για αυτές τις αποστολές. Καταρχήν θέλω να καλώσω την Ντονατέλα στην ε, γραμματεία την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη συνεδρίαση, ήπιαμε ένα ποτό, γιατί η προηγούμενη συνεργατη μας μας ε, εγκατέλειψε μετά από πολλά χρόνια. Είμαστε λοιπόν πολύ ευτυχείς που η Ντονατέλα έγινε μέλος της γραμματείας. Νομίζω ότι την ξέρετε καθότι ήταν στους σοσιαλιστές Είμαι πολύ ευτυχή που την έχουμε μαζί μας, είναι πολύ αποτελεσματική, έχει ήδη ξεκινήσει να δουλεύει και θα ήθελα για άλλη μια φορά να την καλωσορίσω, αν και οι περισσότεροι τη γνωρίζετε. Τι άλλο ήθελα να πω. Αύριο το πρωί με έχουν καλέσει για την άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου για θέματα ανάπτυξης. Με έχουν καλέσει, πρόκειται για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των στόχων θα είμαι βεβαίως εδώ πίσω για τις ψηφοφορίες. <coughs> Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση. Αύριο στην αρχή της συνεδρίασης θα με αντικαταστήσει ο Αντιπρόεδρος. Τι άλλο, η επόμενη Τρίτη έχουμε κοινή ακρόαση για το θέμα της πολιτιστικής ε, πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα μέλη θα είναι παρόντα. Εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι παρούσα, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι τόσο σομαρό που είναι σημαντικό να είμαστε παρόντες. Είναι στο 4Q2 την επόμενη Τρίτη στις 5. 6 Μαρτίου. Εξαιρετική συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας είναι μια συνήθη συνεδρίαση, συνήθως ε, στην εβδομάδα των πολιτικών εβδομάδων, των πολιτικών ομάδων, συγγνώμη, γίνεται μια τέτοια εξαιρετική συνεδρίαση. 8.30 το πρωί. 8.30 το πρωί με 10.30 συνάδελφοι στις 6 Μαρτίου σημειώστε το παρακαλώ και αν μπορείτε να υπενθυμίζετε και στους συναδέλφους. Επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό, διότι και πάλι θα μιλήσουμε για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, αξιολόγηση και θα είναι παρόντες και οι συγητές, αλλά και οι σκιώδεις. από την τελευταία εβδομάδα που ήμασταν σε αποστολές την ε, Πράσινη Εβδομάδα έχουν προκύψει θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των ε, ΜΚΟ. Ξέρετε, τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα για την Oxfam, δηλαδή συνεργάτες της Oxfam οι οποίοι συμπεριφέρονταν με έναν ε, άπρεπο τρόπο, άτομα τα οποία έπαψαν ε, να είναι συνεργάτες της Oxfam αφού αποκαλύφθηκαν όλα αυτά τα γεγονότα. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, έχουν προκαλέσει μια πολύ έντονη συζήτηση όλη την ε, προηγούμενη εβδομάδα και πιστεύω ότι μόλις έχουμε όλα τα στοιχεία και πλήρη ενημέρωση για αυτό που συνέβη, θα πρέπει να το συζητήσουμε εδώ στην ε, συνεδρίαση. Η Επιτροπή νομίζω ότι θα μας ενημερώσει Ξέρω ότι η Επιτροπή έχει ήδη κάνει κάποιες ε, δηλώσεις, κάποιες ανακοινώσεις για το θέμα της Oxfam και θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να μας ε, πει τι ακριβώς ε, έχει αναλάβει σαν δράση μέχρι τώρα. Στο σημείο 6 θα μας δώσει τις πληροφορίες αυτές η Επιτροπή και θα ακολουθήσει βεβαίως συζήτηση όταν είμαστε πλήρως ενημερωμένοι. Έχετε τα πρακτικά της συνεδρίασης 4 Δεκεμβρίου. Μέχρι το τέλος συνεδρίασής μας, παρακαλώ πολύ, αν έχετε παρατηρήσεις, υποβάλλετε τις στην γραμματεία, αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Το ίδιο και για την 24η Ιανουαρίου. Μέχρι το τέλος συνεδρίασης, παρακαλώ πολύ, υποβάλλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, αλλιώς τα πρακτικά της 24 Ιανουαρίου είναι εγκεκριμένα. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της Oxfam, δίνω αμέσως το λόγο στην Επιτροπή, ο Κάρστεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, επιτρέψτε μου να πω μερικά πράγματα για τη δημόσια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τώρα, η οποία ήταν πάρα πολύ σαφής ε, και απλή. Αυτή που, αυτό που έχουμε πει μέχρι τώρα είναι ότι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συνάδουν ε, οι, ε, οι εταίροι της με ηθική και δεοντολογία για οποιασδήποτε λοιπόν ισχυρισμούς σε σχέση με τη χρηματοδότηση των συνεργατών μας. Περιμένουμε να οι ισχυρισμοί αυτοί να διαλευκανθούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης, χρειαζόμαστε περισσότερη επιβεβαίωση ότι η Oxfam μπορεί ως συνεργάτης μας ε, να ε, εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και να τηρήσει τα, ε, τις ηθικές και δεοντολογικές της υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο των μηχανισμών συνεργασίας μας έχουμε ζητήσει λοιπόν να διαλευκαθούν οι ισχυρισμοί αυτοί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και θα γίνουν και πολλές συναντήσεις προκειμένου να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες. Όσο όμως αυτό παραμένει ακόμη εκρεμές, εμείς δεν θα υπογράψουμε περαιτέρω ε, συμφωνίες ανάπτυξης με την ε, Oxfam ε, και επίσης έχουμε αποστείλει στους όλους τους οργανισμούς ε, ε, σαν την Oxfam με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να τους υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και ε, θα γίνεται αναθεώρηση ή διακοπή της χρηματοδότησης αν δεν ανταποκρίνεται κάποιος στις υψηλές ηθικές και διοντολογικές προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνονται στις συμφωνίες μας με τους εταίρους μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δήλωση αυτή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ σήμερα τη απουσία των πληροφοριών για τις οποίες εσείς ε, θέλετε περισσότερες διευκρινήσεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να επενέσουμε ε, το, η δουλειά των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ο Νόρμπερτ και εγώ είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα σε σχετική αποστολή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να δουλεύει κανείς υπό τόσο δύσκολες συνθήκες. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εργασίας. Η Oxfam πάει σε περιοχές στις οποίες, στις εμείς, στις οποίες εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε καν για λόγους ασφαλείας. Οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, να μην ε, δίνουμε την εντύπωση ότι συλλήβδιν καταδικάζουμε όλους αυτούς τους ε, ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που σε αυτές τις ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Οπότε θα γίνει μια συζήτηση, αλλά όχι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τη δήλωση αυτή. Υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Πολύ ωραία. Μπορούμε να κλείσουμε το 6 και να πάμε στο 7, που είναι η δημόσια ακρόαση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θα φύγω από την Προεδρία και θα την παραχωρήσω στον Bogdan Βέντα και στον Βενσό Πεγιό ε, που θα είναι και οι συντονιστές μας για τη σημερινή συνεδρίαση. Δεν θα, κάνω, λοιπόν, την εισαγω... ήθελα λοιπόν να κάνω την εισαγωγή για το σημείο 7 τη ημερήσια διαταξή μα, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Επιτροπή μα ε, και για την εφαρμογή των στόχων ε, αηφόρου ανάπτυξη. Ε, η εκπαίδευση είναι και ένα από τα κέρια σημεία των στόχων, των αναπτυξιακών στόχων τη χιλιετίας και ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών ε, που ενεγράφησαν στα σχολεία κατά την περίοδο 2000-2015, παρά το γεγονός ε, ότι πριν από 18 χρόνια ασκήσαμε τόση πίεση, βλέπουμε τώρα μείωση ε, στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και στο κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση. Είμαι βέβαιη ότι θα ακούσουμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, των παρουσιάσεων για το θέμα αυτό. Πάντως το 2009 10% της αναπτυξιακής βοήθειας αφορούσε την εκπαίδευση εκπαίδευση και τώρα είναι 7%. Ε, στις αρχές του μήνα υπήρξε μία, μία συνάντηση της Παγκόσμιας εταιρική Σχέσης για την εκπαίδευση που είναι ο μοναδικός μηχανισμός χρηματοδότησης ε, για την εκπαίδευση και έλαβε χώρα στο Ντακάρ. Ε, δύο δις συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο αυτού του GPE, της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Εκπαίδευση, για τα επόμενα τρία χρόνια και οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, επίσης ε, είπαν ότι θα διαθέσουν 30 ε, δισεκατομμύρια, όμως πολλές φορές γίνονται τέτοιου είδους υποσχέσεις που τελικά δεν εκπληρώνονται. 110 λοιπόν λοιπόν είναι πλέον τώρα ο προϋπολογισμός μας. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δεν είναι το μόνο πράγμα που είναι σημαντικό η εγγραφή στο σχολείο. Γιατί στην Αφρική, για παράδειγμα, ε, ή μας είπαν ότι υπάρχουν περίπου 160 παιδιά σε κάθε τάξη ε, σε πολλές αφρικανικές χώρες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ε, έλλειψη διδασκόντων και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της, των αναλφαβήτων είναι ενήλικες. 23% ε, μάλιστα των αναλφαβήτων είναι οι γυναίκες. Ε, είναι λοιπόν ε, αυτό πολύ σημαντικό ζήτημα. Σημαντικό είναι και το θέμα των παιδιών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες ή σε ζώνες κρίσεων. Είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να εξετάσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια στην εκπαίδευση και είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο υπαριθμών 4 του, των στόχων αηφόρου ανάπτυξης. Πόγδαν, να σου δώσω το λόγο. Έμεινε στη Σενεγάλη όλο το Σαββατοκύριακο, έμεινε εκεί πέρα καθυλωμένο, είχε δύσκολο Σαββατοκύριο. Όμω ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα, είσαι πολύ αφοσιωμένο ε, ε, στο ε, σκοπό μα. Εγώ θα φύγω, θα σου αφήσω την Προεδρία, θα πάω να κάτσω απέναντι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας ακρόαση. Ε, καλησπέρα, συνάδελφοι, και όπως υπόθηκε ήδη, ε, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος στην ενίσχυση και την προώθηση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Ειδικότερα με την έγκριση των στόχων του υπαριθμού 4, του υπαριθμού 4 για παράδειγμα, που ζητά ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, διαβίου εκμάθηση για όλους μέχρι το 2030 ε, και η εστίαση επεκτείνεται. Δηλαδή δεν αφορά μόνο την, ε, το δημοτικό σχολείο, αφορά και τη δευτεροβάθμια και τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη παροχής δεξιοτήτων ε, και ευκαιριών για απασχόληση ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί στο επόμενο πάνελ μας και επίσης να υπάρξει μία περιεκτική, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλους και διαφύγω εκμάθηση από την προσχολική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή. Ε, ακόμη πιο σημαντικό πρέπει να δούμε την εκπαίδευση όχι μόνο σε ποσοτικούς όρους, αλλά και σε ποιοτικού όρους. Δεν είναι μόνο σημαντικό να αυξήσουμε τον, το ποσοστό εγγραφή στα σχολεία, αλλά πρέπει ε, η σχολική εκπαίδευση να οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα θετικό ως προς την εκμάθηση. Σήμερα το απόγευμα θα ασχοληθούμε με αυτό το ε, συγκεκριμένο σενάριο των στόχων αηφόρου ανάπτυξη διασμού με την εκπαίδευση και ειδικά με τον υπαριθμό 4 ε, στόχο και έχουμε εδώ πολύ ε, εξέχουσες προσωπικότητες, ε, η Άννα ε, Διάτζιο που είναι η οποία είναι η πρώτη μας προσκεκλημένη και είναι υπεύθυνη της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης του 2018 που κατήρτισε η UNESCO, είναι αναλήτρια πολιτικής Η έκθεση αυτή αφορά στη λογοδοσία σε θέματα εκπαίδευσης και αναλύει το πώς μπορούν οι φορείς να παρέχουν πιο αποτελεσματική και πιο επαρκή, ε, πιο επαρκή και πιο ισότιμη εκπαίδευση. Ε, ο μηχανισμός κάλυπτε ολόκληρη την κοινότητα τη σχολική, τους διδάσκοντες, τους γονείς, ε, όλους όσους θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκπαίδευση και να έχουν ένα αποτέλεσμα για την ποιοτική εκπαίδευση. Επί τη βάση αυτών των στοιχείων γίνονται σημαντικές συστάσεις στο πλαίσιο τη έκθεση για το πώ μπορεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο σύστημα εκπαίδευση. Κατόπιν αυτής επισκόπησης της παγκόσμιας κατάστασης, ε, στη δεύτερη, η δεύτερη μα ομιλήτρια ε, θα φέρει πιο κοντά μα το θέμα τη εκπαίδευση. Τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εκπαίδευση στι ε, αναπτυσσόμενε χώρε. Η κυρία Ματέιτσεκ είναι τμήματάρχη στην Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα θέματα εκπαίδευση πολιτισμού και υγεία για θα μας κάνει μια επισκόπηση των ε, προτεραιοτήτων συνεργασίας σε σχέση με την ανάπτυξη ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα μας μιλήσει για τις κατευθυντήριες αρχές αναπτυξιακής πολιτικής, όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θέλουμε να ακούσουμε επίσης περισσότερα ε, για την, ε, τις υπάρχουσες οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με, διαμέσου των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί τα απαιτούμενα αποτελέσματα. μπορεί να έχετε δει ότι υπάρχει ένας ακόμη, ένας κανονικά σε αυτό το πάνελ ο Ντέον Φίλμερ ή Χάλσι Ρότζες, ένας από τους δύο, ε, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στο σημερινό μας πάνελ. Παρ' όλα αυτά, οι δύο μιλήτριές μας θα μας δώσουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα του πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με το στόχο 4 και με την ενίσχυση της εκπαίδευσης. Να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Ντάντιο. Έχετε 10 λεπτά για να μας δώσετε πολλές πληροφορίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ονομάζομαι Ανανταντία και είμαι ανώτερη αναλυτής πολιτικής για την ε, έκθεση της UNESCO για την ε, εκπαίδευση. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε σε αυτήν την κρόση τώρα που τα, ε, είναι πολύ σημαντικές οι στιγμές γιατί θα κάνουμε στην επόμενη περίοδο εκταμιεύσεων. Θα σας εξηγήσω τα της έκθεσής μας, να σας πω τα πιο σημαντικά αποτελέσματα ε, από όσο έχουμε να αναφέρουμε και τι μπορεί να γίνει χρηματοοικονομικά ούτως ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Ένωση στη διεθνή σκηνή. Όπως γνωρίζετε, ο τέταρτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης αποτελείται από τέσσερις στόχους και τρία εργαλεία υλοποίησης και πρέπει όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί το 2030. Θα δείτε αυτά στην παρουσίασή μου και υπάρχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά τις χώρες που καλύπτονται όσον αφορά τις δεξιότητες, όσον αφορά την ισόβια κατάρτιση και αυτή η έκθεση για την εκπαίδευση ε, ξεκίνησε το 2002 και από τότε έχουμε ένα επιτελείο ανεξάρτητο που την ε, συγγράφει και δημοσίευση γίνεται από την ε, UNESCO. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανακατεύεται. Και είναι ένα πείραμα πετυχημένο, γιατί στο Παγκόσμιο την Εκδέση του 2015 πήραμε την εντολή να είμαστε ο μηχανισμός για να αναφέρουμε σχετικά με τα SDG 4 και επίσης για να υποβάλουμε εκθέσεις όσον αφορά τις ε, εθνικές και όχι μόνο στρατηγικές για όλους τους εταίρους μας όσον αφορά την εκπαίδευση. Οπότε και το αποτέλεσμα αυτής της διτής εντολής ήταν ότι η έκθεση έχει δύο τμήματα. Το ένα τμήμα αφορά το υποπτικό κομμάτι για τους στόχους αυτούς που αναφέραμε προηγουμένως και υπάρχει και το θεματικό τμήμα που αφορά τις μελέτες που γίνουν από τους συμβούλους μας. Το 2016 έχουμε τα θέματα παιδείας και τους άλλους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης. Μετά έχουμε την ε, λογοδοσία Στη συνέχεια το 19 θα έχουμε ε, βασικό θέμα την μετανάστευση και τον εκτοπισμό ή τη μετακίνηση και την ένταξη το 20. Να σας πω επίσης τι γίνεται με τους στόχους που καλύπτουμε στην εκθεσή μας. Πρώτα πρώτα έχουμε τον στόχο 4.1. Να δούμε τι πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά για την υποχρεωτική και ποιοτική παιδεία. Έχουμε 264 εκατομμύρια παιδιά, ακόμη είναι εκτός σχολείου. Οπότε το να πάει κανείς σχολείο δεν σημαίνει ότι θα αποφυτίσει. Επίσης την περίοδο 10 με 15 είχαμε 83% που αποφύτησαν από το δημοτικό, 60 για τη δευτεροβάθμια και 40 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε εδώ μπορείτε να δείτε πώς γίνεται η κατανομή ε, ανά χώρα. Το ποσοστό ήταν 83, 69 για δευτεροβάθμια και 45 για το πανεπιστήμιο. Ε, αυτή η κατάταξη έχει γίνει σύμφωνα με τους ρυθμούς ε, Και βλέπετε σχετικά εδώ τις πράσινες τελίτσες. Και έχουμε τις διαφορές χώρα Οπότε μπορείτε να διαπιστώσετε ότι έχουμε τουλάχιστον 15 χώρες στα αριστερά της γραφικής παράστασης, εκεί που είναι οι μπλε κουκίδες και εκεί έχουμε λιγότερα από ένα ε, παιδί, λιγότερο από ένα παιδί που αποφύτησε στην από την πρωτοβαθμία παιδεία. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο η αποφύτιση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει σε μαθηματικά και ανάγνωση ε, ποιοτική εκπαίδευση. Δεν έχουμε κάποιο είδου ενιαία στάνταρ για αυτά, αλλά έχουμε προχωρήσει όσον αφορά την Παγκόσμια Συμμαχία Παρακολούθησης της εκπαίδευσης και έχουμε την έκθεση του 12, οπότε και το Ίδρυμα Σταστικών της UNESCO υπολόγισε ότι ένα στα δύο παιδιά που αποφυτούν από το δημοτικό δεν έχει αυτές τις βασικές ικανότητες, δηλαδή να ξέρει μαθηματικά και ανάγνωση. Και πράγματα είναι 9 στα 10 στην Αφρική νοτίου της Σαχαράς. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει ε, να διαπιστώσουμε ότι λιγότερο από μία πέντε χώρες έχουν εγγύσεις ε, για 12 ετή υποχρεωτική παιδεία. Λιγότερε από μία στις πέντε. Τώρα, στόχος 4, 2. Εδώ έχουμε τα θεμέλια για την γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει γενική συμφωνία για τον ορισμό σε σχέση με το σχολείο. 69% ε, σύμφωνα με τη στατιστική της UNESCO 69% ήταν τα παιδιά που σκότωσαν στο σχολείο στην ε, ηλικία που είναι πριν από αυτήν που προβλέπεται. Ε, αλλά βέβαια πολύ χειρότερα τα πράγματα στην Καραϊβική και στην ε, Αφρική νοτίως της ε, Σαχάρας. Επομένω βλέπουμε ότι ε, έχουν χάσει το τρένο αυτοί οι μη προνομιούχοι. Και το 2010 2015 τα πιο πλούσια παιδιά είχαν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να πάνε σε σχολείο από ότι τα πιο φτωχά και τα παιδιά από αστικές περιοχές είχαν διπλάσιες πιθανότητες ούτως ώστε να πάνε ε, στο σχολείο σε σχέση με τα παιδιά που ζουν στην Ήπεθρο. Οπότε βλέπουμε, σύμφωνα με το πώς γράφεται στο σχολείο, ότι υπάρχει πρόοδος. Αλλά μόνο 17% των ε, χωρών έχουν ε, νομική ρύθμιση όσον αφορά την υποχρεωτικότητα ε, για την ε, περίοδο της εκπαίδευσης πριν το δημοτικό. Να δούμε τώρα τον χάρτη 4-5 ε, γιατί εδώ πέρα το θεματολόγιο μας οδήγησε σε μια σημαντική στροφή για να μην χάσει κανείς πια το τρένο. Και είπαμε ότι στον στόχο 4,5 καλυπτόμαστε όσον αφορά αυτού του είδους την δικαιοσύνη στην παιδεία. Τι γίνεται τώρα. Διαφέρει κατάσταση αναπίπεδο παιδείας και αναχώρα μόνο 60% των χωρών έχουν ε, πετύχει αυτήν την ισότητα. 45% σε δεύτερο βάθμια ε, και 50% για την ε, ανώτερη βάθμια παιδεία. Βλέπετε εδώ σε αυτό το διάγραμμα τι ισχύει όσον αφορά τις πληροφορίες μας για την ισότητα στην παιδεία και βλέπετε εδώ πέρα ποια είναι τα κενά και οι ανισότητες. Ας πούμε, στο Σαλβαδόρ έχουμε 51% των πιο πλουσίων, αλλά λιγότερο από 2% ε, των ε, πιο φτωχών συνέχισαν την εκπαίδευση μετά τη δευτεροβάθμια φάση. Στη Μογγολία επίσης έχουμε 67% και 3% αντιστοίχως επίσης από την έκθεση προκύπτει το πώς καταγράφονται. Αυτές οι ανισότητες. Ένα στα εκατό φτωχά κορίτσια φίδησαν σε σχολείο. Αλλά βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει υποτίμηση των ανισοτήτων και οι πιο ευάλωτοι είναι αυτοί που έχουν ευκαιριακές, εποχιακές δουλειές, οι άστεγοι και αυτοί όλοι δεν καλύπτονται από τις ε, έρευνες για τον τρόπο που είναι φτιαγμένες. Και έχουμε 250 εκατομμύρια που δεν καλύπτονται λόγω της μεθοδολογίας των ερευνών. Πάμε τώρα στον στόχο 4α όσον αφορά το μαθησιακό περιβάλλον. Βασίζεται στην αρχή ενός σχολείου φιλικό στα παιδιά. Άρα εδώ είναι και το θέμα οι υποδομές αλλά και η βία στο σχολείο. Δύσκολο, δύσκολο να έχουμε όμως με την πλήρη εικόνα. Ενδεικτικά όμως, ξέρουμε ότι στην Αφρική, νοτιού της Σαχάρας, τα 4 πέμπτα των πρωτοβαθμίων σχολείων δεν έχουν ηλεκτρισμό και σε όλο τον κόσμο το 1 τέταρτον των δημοτικών σχολείων δεν έχουν πόσιμο νερό. Επίσης, οι μελέτες και έρευνα σαν ανεδεικνύουν το ότι υπάρχει πρόβλημα με την υποδομή. Και αυτό είναι κάτι που έχει σχέση βέβαια με τον πλούτο κάθε χώρας και τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα στις ε, μη προνομίχες περιοχές. Επίσης, έχουμε το θέμα των επιθέσεων έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις στα σχολεία από το 2004 σε Νότια Ασία, Βόρεια Αφρική και στη Δυτική Ασία, πολύ περισσότερο από διαλόγου και στην Ιγυρία έχουμε 19.000 δασκάλων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα μεταξύ 2009 και 2015. Το 2016 στην Συρία είχαμε πάνω από τον τέταρτον των σχολείων που καταστράφηκαν. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο σημαντικό. Ο στόχος 4C που αφορά την προσφορά σε δασκάλους που έχουν σωστές δεξιότητες, που το 86% έχουν εκπαιδευτεί για το ε, δημοτικό, αλλά βλέπουμε ε, ότι διαφέρει ανά Ασία το ποσοστό 60% στην Αφρική, 70% στην Καραδική και στην Ασία. Βλέπουμε όμως ότι είναι παραπλανητική αυτή η σύγκριση γιατί έχουμε πάρα πολλές διαφορές που δεν έχουν καταγραφεί όσον αφορά τα ελάχιστα προαπαιτούμενα ούτως ώστε να χαρακτηριστούν το ποιοι είναι οι δάσκαλοι που έχουν αυτά τα προσόντα, τις δεξιότητες, για το βιογραφικό τους, ε, το, το, το χρόνο εκπαίδευσή του κλπ. Υπάρχει πάντως μια θετική στάση όσον αφορά τους εκπαιδευμένου δάσκαλου σε κάποιες χώρες νοτίω τη Σαχάρα τη Αφρικής και βλέπουμε εδώ τα στοιχεία ότι ιδίω σε Ερυθρέα, Νίγηρα και Γκάνα. Το σχετικό ποσοστό των εκπαιδευμένων δασκάλων συρρυκνώνεται από το 2000 και αυτό λόγω της ε, αύξησης των προσλήψεων συμβασιούχων δασκάλων που έχουν όμως χαμηλές δεξιότητες και προσόντα. Όσον αφορά τα κίνητρα για τους δασκάλους, δηλαδή σε σχέση με την ε, ε πρόοδό τους, την καριέρα τους ε, και λοιπά, του το αν κουράζουν τη δουλειά. Βλέπουμε δύο σε χώρες του ΩΣΑ ότι οι δάσκαλοι στα δημοτικά κερδίζουν 81% από όσο άλλοι εργαζόμενοι που έχουν ιδίου επίπεδου πτυχία. Για να δούμε τώρα τα θέματα τα χρηματοοικονομικά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό σημείο υλοποίηση της ε, πολιτικής μας. Ακόμα και αν αυτό δεν έχει περιληφθεί στο SDG 4, έχει σχέση όμως με αυτό το εξαζόμενο πλαίσιο όσον αφορά τι δημόσιε δαπάνε. Μία στι τέσσερι χώρε δεν μπόρεσε να καλύψει τα κριτήρια για να ξοδεύει, για να έχει 4% του ΕΠ ή 15% του προπολογισμού. Και όσον αφορά τις ενισχύσεις, μόνο 6 από 28 δωρητέ ετήρησαν το 0,7% του να δώσουν στις ενισχύσεις αυτό το ποστό από το ΑΕΠ τους. 10% επομένως αυτής της ε, ενίσχυσης πήγε σε δημοτικά γυμνάσια, αλλά ε, μειώθηκε το σύνολο. Ε, μειώθηκε μέσα σε μια εξαετία κάθε χρόνο και συνέχεια έπεσε περίπου στο 7% το οποίο είναι 4% λιγότερο σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα την περίοδο 9 έως 10. Στην έκθεσή μας πολλά χρόνια έχουμε αναδείξει ότι οι κυβερνήσεις και οι δωρητές καλύπτουν μόνο τμήμα του κόστους. <coughs> Στις δε πλούτιες χώρες οι δαπάνες καλύπτονται από τις οικογένειες. Και στις πιο φτωχές χώρες έχουμε 33% που καλύπτουν. Και σε κάποιες χώρες όπως την Καμπότζη είχαμε 61% που καλύπτεται από τις οικογένειες. Γι' αυτό βλέπετε στην γραφική παράσταση στην Καμπότζη στην Άκρη, άκρη. Για να δούμε τώρα. Έχουμε και τις γραφικέ γραφικές παραστάσεις όσον αφορά την ε, ενίσχυση στην παιδεία. Έχουμε αυτό το έγγραφο για την πολιτική μας και δείχνει τα στοιχεία του ΩΣΑ και διαπιστώνεται από αυτά τα στοιχεία ότι η ενίσχυση για την εκπαίδευση έχει βαλτώσει, είναι σε στασιμότητα την περίοδο 9-10 στο ποσό των 12 δις δολαρίων και περίπου 5 δις διατίθενται για την βασική εκπαίδευση, αλλά μόλις 1,3 δις πηγαίνουν στην Αφρική και επομένως ε, τώρα παίρνει τα μισά λεφτά η Αφρική από όσο έπαιρνε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000. Επίσης έχουμε κάποιο είδους διμερείς δωρεές που εκταμιεύουν 62% του συνόλου της ενίσχυσης αλλά οι πολυμερείς αύξησαν το μεριδιό. Πάμε παρακάτω τώρα. Ε, τα επόμενα στοιχεία μας δείχνουν την εξέλιξη των ενισχύσεων για τη βασική εκπαίδευση σε σχέση με τα πέντε πολυμερή θεσμικά όργανα και βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος πιο μεγάλος χρηματοδότης για τη βασική εκπαίδευση. Και αυτά τα επίπεδα είναι σταθερά για την Ένωση από το 2005, περίπου στα 5 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά υπάρχει αυξητική τάση μεταξύ 2013 και 2016, γιατί πήγαμε στα 500 εκατομμύρια. Για να δούμε τώρα την τελευταία διαφάνεια. Εδώ καλύπτουμε το θέμα της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την εκπαίδευση GPE είναι οι υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δόθηκαν στο Ντακάρ και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Εδώ βλέπετε πως έχει εξελιχθεί αυτή η ενίσχυση του GP και μέχρι το 2015 είχαμε 450 περίπου εκατομμύρια ετησίως και σε σχέση με τη στασιμότητα άλλων ενισχύσεων έχουν αυξηθεί τα ποσά του GP 6-12% 2012-2015 για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και άρα πάμε για μεγαλύτερη αύξηση με το 2020. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η ενίσχυση καλύτερα λειτουργεί όσον αφορά τις πιο φτωχές χώρες σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα για την παιδεία. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί έκανα λάθος στην αρχή. Αλλά και τώρα έχουμε άλλα 10 λεπτά για την επόμενη παρουσίαση για να μας μείνει χρόνος για συζήτηση και απάντηση σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την Agenda 2030, Καταρχήν θα ήθελα να επανέλθω στις βασικές μας προκλήσεις. Όλες οι γενικές διευθύνσεις ε, έχουν ε, ένα κοινό στόχο πώς θα βελτιωθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Βεβαίως η DG το είναι αυτή που έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο Όσον αφορά το SDG 8 και το 4, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου κάποιους αριθμούς. 260 εκατομμύρια παιδιά και νέοι δεν πηγαίνουν σχολείο και δεν έχουν καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα επίσης και με κάποια παιδιά που ναι μεν βρίσκονται στα σχολεία αλλά δεν έχουν καθηγητές, δεν έχουν δασκάλους. 68,8 εκατομμύρια δάσκαλοι. Είναι τα νούμερα που έχουμε για το 2018 λοιπόν κατάσταση επίσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Τα κορίτσια πηγαίνουν πολύ λιγότερο στο σχολείο από τα αγόρια. Βεβαίως και το θέμα των εκτοπιστέντων, των κρίσεων, των ανθρωπιστικών κρίσεων. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις πατρίδες τους, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, πλήττονται άμεσα από το θέμα αυτό της ε, εκπαίδευσης και της κατάρτισης και τουλάχιστον 30 εκατομμύρια παιδιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός ε, των περιοχών όπου θα μπορούσαν να πάνε στο σχολείο ή να έχουν κάποιο άλλο είδους εκπαίδευση ή κατάρτιση. Βεβαίως ε, τα προβλήματα που ακολουθούν είναι γνωστά. Πέρα από την χρηματοδότηση, πέρα από την δημιουργία σχολείων, έχουμε θέσει βασικές προτεραιότητες. Ενσωμάτωση των φίλων, η εκπροσώπηση και αυτό σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης μέχρι και την ανώτατη. Το θέμα των ε, καθηγητών, των δασκάλων, το θέμα των ε, περιοχών ε, όπου επικρατούν δύσκολες συνθήκες κρίσεις και βεβαίως το θέμα της απασχολησιμότητας της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας των νέων. Εργαζόμαστε σε τρία επίπεδα. Διμερής στήριξη, περιφερειακά προγράμματα και οι προτεραιότητες οι οποίες ονομάζονται Global Initiatives Όσον αφορά τις ε, διμερείς ε, βοήθειες και τα προγράμματα διμερού συνεργασίας, 49 χώρες συμμετέχουν. Συμμετέχουν επίσης ιδιωτικές επιχειρήσεις για τις ε, περιφερειακές ε, αυτές ε, πρωτοβουλίες και προγράμματα. Έχουμε τρεις τομείς, τους οποίους δραστηριοποιούμαστε, το Erasmus Plus, ανταλλαγές μεταξύ ανθρώπων, διαπολιτισμικός διάλογος και φυσικά ο εξυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης. Erasmus Plus που έχει μία παγκόσμια διάσταση ξεκίνησε ήδη από το 2014 έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε κοινά μάστερ, σε προγράμματα κοινής εκπαίδευσης πάνω από 150 Και βεβαίως ο δεύτερος τομέας στον οποίο δραστηριοποιούμαστε σε περιφερειακό επίπεδο με περιφερειακά προγράμματα είναι το επίπεδο DCI. Πρόσβαση στην παιδεία, στην εκπαίδευση, σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση, η κατανόηση δηλαδή των νέων αυτών εργαλείων ποια είναι αυτά που μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε περίοδο κρίσης. Προγράμματα DCI που έχουν ξεπεράσει φέτος το 2018 όσον αφορά τις δεσμεύσεις τα 20 εκατομμύρια. ΒΕΤ σε περιφερειακό πάντα επίπεδο με την συνεργασία σημαντικών φορέων όπως το British Council και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, προσφορά δηλαδή στήριξης, κατάρτισης, τεχνογνωσίας υψηλού επίπεδου, ενίσχυση της δράσης των φορέων του ιδιωτικού τομέα. Προσπαθούμε δηλαδή να ενσωματώσουμε όλο και περισσότερους φορείς του ιδιωτικού τομέα ε, στα διαφορετικά ΒΕΤ. Όπως είπε η κυρία Ντάντιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος ε, χρηματοδότης. Έχουμε ήδη προσφέρει πάνω από 300 εκατομμύρια και άλλα 100, 175 μέχρι το 2020 για τη διετία 18-20. Είναι η μοναδική ολοκληρωμένη εταιρική σχέση που έχει στο επίκεντρό της την ε, εκπαίδευση όλων των ε, επιπέδων με τρεις πολύ σημαντικούς στόχους. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την όθηση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων. Να στηρίξουμε τις GPE, να βοηθήσουμε τους καθηγητές, να στηρίξουμε τα προγράμματα κατάρτισης καθηγητών και εκπαιδευτικού προσωπικού και βεβαίως ε, να στοχεύσουμε και να ενσωματώσουμε και τους πιο περιθωριοποιημένους, τις πιο ευάλωτες ομάδες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά μας σε επίπεδο περιφερειών. Για το 2018 έχουμε 89 αναπτυσσόμενες χώρες και στοχεύουμε 870 εκατομμύρια παιδιά και νέους. Αυτά προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. 19 εκατομμύρια επιπλέον παιδιά τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση, το δημοτικό, και πάνω από 10,8 παιδιά τα οποία βρίσκονται σε χώρες με σειράξεις, συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις. 1,7 εκατομμύρια καθηγητών έχουν ε, περάσει από σεμινάρια κατάρτισης και έχουν ολοκληρώσει την κατάρτισή τους σε 23.800 σχολεία, αίθουσες σχολικές, 204 εκατομμύρια εγχειρίδια, σχολικά βιβλία έχουν μοιραστεί για το 2017. Το 2002, συγγνώμη, το 2014 διορθώνει η ομιλήτρια, 64 εκατομμύρια παιδιά μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τάξεις και τα σχολεία του Δημοτικού σε σχέση με το 2002 δηλαδή συν 64 εκατομμύρια. Και το 73% των παιδιών ε, αυτών ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας βασικός, ε, αν θέλετε, στόχος μας είναι να περάσει το μήνυμα ότι η εκπαίδευση, η παιδεία, η κατάρτιση δεν είναι κάτι που μπορεί να αναβληθεί και είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι οι στόχοι μας υλοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα σε στρατόπεδα προσφύγων. Το 2017 έχουμε καλύψει την εκπαίδευση 4 εκατομμύριων παιδιών και νέων, ιδιαίτερα μετατοπιστέντων προσφύγων σε 14 διαφορετικές περιοχές που πλήττονται από κρίση, από σειράξεις και σε στρατόπεδα μεταναστών και προσφύγων. Έχουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες που όπως είπα δεν μπορούν να περιμένουν, δεν μπορούν να αναβληθούν, πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Υψηλής ποιότητας προσφορά κατάρτισης, ανθρωπιστική, επιπλέον δηλαδή της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσφέρουμε στα στρατόπεδα των προσφύγων. Τέλος, Θέλω να πω δύο λόγια για το IFED. Φαντάζομαι γνωρίζετε την πρωτοβουλία αυτή που είναι η διεθνής χρηματοδότηση προς ε, τις πρωτοβουλίες αυτές εκπαίδευσης. Παρακολουθούμε στενά τις ε, συστάσεις που έχει υποβάλει η Επιτροπή για την ε, Παιδεία και την Εκπαίδευση Βεβαίως και περιμένουμε να λειτουργήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν κενά στις χώρες όσον αφορά την χρηματοδότηση των συστημάτων αυτών. Να μην αφήσουμε δηλαδή καμία χώρα με κενά όσον αφορά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Γι' αυτό και στηρίζουμε και παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή την ε, νομική προετοιμασία, το νομικό πλαίσιο των ε, χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων που έχουν σαν σκοπό να στηρίξουν τα προγράμματα αυτά, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες χώρες. Αυτή είναι η πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Ε, τώρα θα αρχίσει η συζήτηση. Παρακαλώ να συστηθείτε πρώτα και μετά να θέσετε την ερώτηση στους κύριους Πεγιών πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, γίνεται μία διάγνωση της κατάστασης. Ε, το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω για να κατανοήσω καλύτερα. Υπάρχει πρόοδος, αλλά είναι λιγότερα τα χρήματα, αν κατάλαβα καλά. Το να ζητήσουμε όμως περισσότερα χρήματα με βάση αυτή την επιχειρηματολογία δεν τα καταφέρουμε. Δηλαδή υπάρχει πρόοδος ενώ μειώνεται η χρηματοδότηση, υπάρχει μια μικρή δυσκολία. Τι δικαιολογεί κατά τη γνώμη σας, πώς εξηγείται αυτή η μείωση της ε, χρηματοδοτικής βοήθειας, όχι σε απόλυτους όρους, αλλά σε σχετικούς όρους. Γιατί επειδή οι χώρες επενδύουν εκείνες περισσότερα χρήματα, είναι επειδή λόγω των κρίσεων ε, ή άλλο, λόγω άλλων τομέων ε, που ε, έχουν προτεραιότητες, κάνουν επενδύσεις πιο μακροχρόνιες. Τι ακριβώς δικαιολογεί αυτό το γεγονός σήμερα. Ε, είπατε ότι αναφερθήκατε στην πρόσφατη σύνοδο του Ντακάρ ε, και είπατε ότι τα ποσά ε, δεν είναι αυτά τα οποία είχαμε φανταστεί. Τρία δις ε, περιμέναμε, δεν τα έχουμε. Εγώ ήμουν ε, κάποτε υπουργό παιδείας στη Γαλλία και το είχαμε αυτό το ε, πρόβλημα. συχνά δεν έχουμε την συγκέντρωση των ποσών που θέλουμε. Λοιπόν, εσείς που είστε λοιπόν οι δήμονες, μήπως μπορείτε να μας πείτε τι, τι, συμβαίνει, για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Η ερώτηση είναι και προς τις δύο σας είναι πάρα πολύ ποσοτική η προσέγγιση Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μια μορφή ε, επιφύλαξης, προσοχής. Μας δίνεται κάποια στοιχεία αριθμητικά τα οποία εμείς δεν τα έχουμε στη θέση μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εγώ θα ήθελα και μια πιο ποιοτική προσέγγιση. Κυρίως όσον αφορά το σχολείο. Γιατί αν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και έχουμε σημειώσει πρόοδο, το είπαμε αυτό ποια είναι τα βασικά εμπόδια, τα εμπόδια των δικών μας των διαδικασιών. Υπάρχει μια πολλαπλότητα παικτών, φορέων κατά την άποψή μου. Ακούσαμε για παράδειγμα ότι σε κάποιες χώρες αναπτυσσόμενες ο συντονισμός δεν είναι πάντοτε ο βέλτιστος λέμε ότι κάνουμε σαν να είναι τυποποιημένη εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ε, επειδή γνωρίζω το εκπαιδευτικό σύστημα και έχω προσπαθήσει να το διαμορφώσω. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Ε, είναι σε μια χώρα της Ευρώπης ε, εύκολο, σε μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολο να τυποποιηθεί κάτι τέτοιο γιατί πολλές χώρες θεωρούν ότι είναι κάτι τέτοιο ένα πολύ εθνικό θέμα. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε, ακόμη και σε αυτά που κάνουμε εμείς, με όλη μας την καλή θέληση, αν υπάρχουν εμπόδια τα οποία πρέπει να αρθούν. Καταρχάς όσον αφορά την πολλαπλότητα των διαφόρων ε, μεθόδων μας, ε, των φορέων μας και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκουμε τις χώρες στις οποίες θέλουμε να βοηθήσουμε. Πρώτον, για πιο λιγο, για λόγο λιγότερα χρήματα και δεύτερον, ε, πιο ποιοτικά ποια είναι τα σημεία όπου το σύστημα αντιμετωπίζει εμπόδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις και θα συνεχίσω ε, αυτά που είπε ο συνάδελφος. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Γνωρίζετε ότι η UNESCO έχει χάσει πολύ μεγάλη χρηματοδότηση φεύγοντας από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, ε, υπάρχει ο στόχος, ο αναπτυξιακός στόχος ε, της εκπαίδευσης για όλους εγώ ήμουν ε, πρέσβυρα τότε, ε, υπάρχουν ακόμη 260 εκατομμύρια παιδιά τα οποία ακόμη δεν ε, πηγαίνουν στο σχολείο και είπατε ότι μόνο 2% της ανθρωπιστικής βοήθειας πηγαίνει στην εκπαίδευση, αν κατάλαβα καλά. Αυτό πραγματικά είναι ιδεχθές. Τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτό το συντονισμό για τον οποίο μιλάμε να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό της αναπτυξιακής βοήθειας, γιατί ε, όταν πηγαίνει κανείς στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, είναι αυτό το πρώτο πράγμα που βλέπει, ότι ε, αν ε, δεν υπάρχουν καν οι εγκαταστάσεις για να πάει κανείς σε σχολείο, δεν μπορεί η χώρα να κάνει και πολλά γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σάχλ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο όταν άκουσα τον Βενσόν ε, θεώρησε ότι δεν μπόρεσα να πω τίποτε το πρωτότυπο μετά από εκείνον. Συμφωνώ λοιπόν με τα σχόλιά του. Όσον αφορά τώρα την ποσοτική ε, προσέγγιση ε, επί της οποίας σχολίασε, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δούμε και τη δημογραφική πτυχή πριν από τη συνάντηση ήρθε ένας εκπρόσωπος της ΦΝΟΑΠ η οποία μόλις είχε μία συνάντηση, μία συνομιλία με τον δήμαρχο του Αμπιτζάν και είπε έχω 300 ε, γεννήσεις την ημέρα. Ε, αν ε, χτίζω ένα σχολείο κάθε μέρα και αν δεν χτίζω ένα πανεπιστήμιο κάθε έξι εβδομάδες, πείτε μου πώς είναι δυνατόν να στεγάσω όλους αυτούς τους μαθητές, τους μελλοντικού μαθητές και φοιτητές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Η δημοκρατική πτυχή είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε στη συζήτησή μας. Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, και αυτό να το λάβουμε υπόψη γιατί μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος Νόρμπερτ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το θέμα που έθεσε ο Σάρλ είναι καθοριστικό, εξαιρετικά σημαντικό. Οι δημοκρατικές, ε, αν θέλετε, εξελίξεις προκαλούν σημαντικά προβλήματα. Βλέπουμε στην υποχασαχάρια περιοχή πώς αυξάνονται οι αριθμοί σε όλους τους ανησυχιστικούς τομείς. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής στην Ευρώπη ήδη λέμε ότι θέλουμε μία δωρεάν εκπαίδευση στην καλύτερη περίπτωση από τον υπιαγωγείο μέχρι το ε, πανεπιστήμιο. Ας ξεκινήσουμε όμως με την κατώτερη, τη βασική εκπαίδευση. Αν μπορούμε να εγγυηθούμε αυτό ήδη, νομίζω ότι κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό και βλέπω ότι πολλά κράτη προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στόχο. Οι στατιστικές όμως και τα στοιχεία που έχουμε είναι εξαιρετικά ε, ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά. Πώς μπορούμε όμως να επηρεάσουμε την πραγματικότητα, αυτό με ενδιαφέρει. Πώς μπορούμε, παραδείγματο χάρη, να κατονομάσουμε και να κατηγορήσουμε τις χώρες αυτές οι οποίες ε, λένε μεν ότι έχουν κάνει πρόοδο, αλλά τίποτα στους τομείς αυτούς που θεωρούμε εμείς τομείς προτεραιότητας. Είναι σημαντικό επίσης εκεί όπου πραγματικά υπάρχει πρόοδος, εκεί που πραγματικά η πρόοδος, η εξέλιξη πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό να αναγνωρίζεται από την κοινότητα και να στηρίζουμε και να βοηθούμε τις χώρες που κάνουν τέτοια θετικά βήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά αριθμητικά στοιχεία ε, ακούσαμε και πέρναγαν πολύ γρήγορα η διαφάνεια. Συγγνώμη λοιπόν να ρωτήσω κάτι που το καλύψατε. Ε, η πρώτη ερώτηση είναι προς την κυρία Ντάντιο. Γιατί ε, είναι ένα πράγμα να έχουμε διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία από διαφορετικές χώρες, αλλά συγκρίνουμε ε, παρόμοια πράγματα, χώρες με παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης και χώρες με παρόμοια επίπεδα ζωής, χώρες που έχουν ε, παρόμοιο επίπεδο ζωής αλλά τα αποτέλεσμα είναι καλύτερο, δεν έχει νόημα την ε, κεντροαφρικανική δημοκρατία να την συγκρίνουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να συγκρίνουμε όμοια πράγματα μεταξύ τους. Αυτό έχει νόημα για να υπάρχει ένα, να, να, να γνωρίζουμε πράγματι πολύ καλά ποιο είναι το αποτέλεσμα για τα παιδιά. Μπορεί κάποιες κυβερνήσεις να κάνουν κάτι ε, από το οποίο μπορεί να μάθουν άλλες ε, ε χώρες. Τουλάχιστον έτσι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και η εκπαίδευσή τους είναι μόνο ένα από τα αποτελέσματα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούμε τις, ε, τα σχολεία ε, ε, και χώρους στους οποίους όπου γίνονται εμβολιασμοί, όπου μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες, όπου κάνουμε μία μέτρηση της κατάστασης υγείας των παιδιών. Στη δική μου χώρα μπορεί να κάνουμε, περισσότερα, να κάνουμε λιγότερα πλέον ε, ως προς τον τομέα της ε, διατροφής των παιδιών, γιατί θεωρούσαμε ε, κάποτε ότι αυτό δεν ήταν ε, ε, ένα καλό στοιχείο των σχολείων μας και τώρα έχουμε υπαναχωρήσει σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν στόχοι που υπερβαίνουν την εκπαίδευση και νομίζω ότι projects στα οποία η UNICEF και άλλες, άλλοι οργανισμοί δίνουν καλλιτικά στις γυναίκες ή παρέχουν διάφορα στοιχεία διάφορα ε, στοιχεία πολύ σημαντικά για τους μαθητές ε, ε, κάνουν πολύ σημαντικό έργο έρχονται από πολύ μακριά για να το κάνουν αυτό ε, υπάρχουν παιδιά που περπατάνε τρία χιλιόμετρα για να πάνε στο δημοτικό σχολείο τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις αυτές. Μας δείξατε και μία διαφάνεια για τις οικογένειες. Ε, πραγματικά είναι σκανδαλώδες ότι όσο φτωχότερος είναι κανείς τόσο περισσότερα πρέπει να πληρώνει. Όταν πήγα στην Αφρική πριν από μερικά χρόνια... Ε, πολλά χρόνια μάλλον, το 2002 στον Γκάνα, όπου κάποιο αξιωματούχος του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου μου, είπαν, μου είπε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια οικονομική εισφορά για τα σχολεία ε, στην ε, Γκάνα, γιατί διαφορετικά δεν θα αξιολογούσε κανείς, δεν θα θεωρούσε πολύτιμα τα σχολεία. Και αυτός ήταν Σουηδό. Μου έκανε εντύπωση αυτό λοιπόν. Ε, εν πάση περιπτώσει αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι Υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι αν πληρώνει κάποιος κάτι, τότε το θεωρεί, πολίτικο, το θεωρεί πολύτιμο. Όχι. Η εκπαίδευση είναι κάτι το πολύτιμο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το πληρώνει κανείς για να το θεωρεί ε, πολύτιμο. Μα είχα δει, με δει μάλιστα και ένα βίντεο, νομίζω για τη Σελεγάλη, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για κάποια παιδιά, για κάποιους νέους για τους οποίους οι γονείς δεν είχαν πληρώσει για τα βιβλία τους και συνεπώς δεν μπόρεσαν να δώσουν εξετάσεις. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα ε, και είναι κάτι το οποίο ανακύπτει συνεχώς όταν επισκεπτόμαστε αυτές τις χώρες. Ε, τα ε, χρήματα που πηγαίνουν στα σχολεία δεν είναι αρκετά οι διδάσκοντες δεν πληρώνονται. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αν δεν πληρώνονται καλά οι δάσκαλοι, ε, ε, τότε ζητούν τις, ε, τις εισφορές των γονέων. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους χώρες σε παρόμοια κατάσταση, οποίες τις συγκρίνεται για να μάθουν η μία από την άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Βέντα. δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, τότε να δώσουμε το λόγο για πέντε λεπτά στην ομιλήτρια τις απαντήσεις. Α, γιατί τη Σενεγάλη. Ναι, ναι, την αναφέραμε δύο φορές. Και εκείνο το καταπίστευμα, εκτό από τα θέματα της παιδείας, μίλησαμε και κατά τη γνώμη μου για την εκπαίδευση. Θα πρέπει να διπλώσουμε ότι έχει η χώρα την απαραίτητη σταθερότητα. Ε, βέβαια, για τα διάφορα προγράμματα είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση. Και η σταθερότητα δεν ισχύει για πολλές χώρες, ιδίω εκείνη την περιοχή του κόσμου. Δύσκολο να βοηθήσει κανείς, δύσκολο κάτι να οργανώσει. Αρκετά σας είπα, εσείς έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις σας. Να σας αναφέρουμε κάποια στοιχεία και μετά να συνεχίσουμε την συζήτηση. Πρώτα-πρώτα. Νομίζω υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία τίθενται τα πρώτα. Διαπιστώθηκε κάποια πρόοδος, αλλά είχε και πάρα πολύ εντυπωσιακή. Επίσης διαπιστώσαμε ότι οι εκταμιεύσεις από τον προϋπολογισμό παραμένουν οι ίδιες ή και βαίνουν μειούμενες. και είπαμε ότι δεν θα υπάρξει πρόοδο στο μέτωπο των παιδιών που καταλήγουν το σχολείο ή που δεν πάνε σχολείο. Είπαμε για το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί όλο ένα και μεγαλώνει ο πληθυσμό της Αφρικής που έχει σημασία. Είναι επομένως δυναμικό το φαινόμενο. Και σε 5-6 χρόνια θα φανούν οι συνέπειες όταν δούμε τι γίνεται στο δημικό, στην πρωτοβάθμια παιδεία. Επομένω, η πληθυσμιακή ομάδα στην οποία αναφερόμαστε θα έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο αύριο. Επίσης, έχουμε φτώχεια εκτεταμένη και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα θέματα της παιδείας. Και φέτος ετοιμάσαμε μια σχετική μελέτη για τις επιπτώσεις του να ξεφύγει κανείς από την παιδεία, να δώσει κανείς παιδεία στον κόσμο, τη βασική παιδεία. Πόσο επομένω στη συνέχεια ξεφεύγει κάποιος από την κατάσταση αυτή. Δεν υπάρχει πρόσβαση στην υγεία, είναι θέματα ακόμα και διατροφής. Αυτοί που έχουν τα πάνε μακριά, κάνουν αποστάσεις για να πάνε στο σχολείο. Και τόσο αυτό το, το θέμα της απόστασης έχει σημασία για την παιδεία, αλλά δεν ανήκει με τη στενή έννοια στην, στο, στο, στο κονδύλι της ε, παιδείας. Επομένω θα πρέπει να τα δούμε σφαιρικά. Α, και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Οι επιπτώσεις των πολέμων που οδηγούν σε μεγάλες μετακίνησει του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. Και δεν μιλώ μόνο για πρόσφυγες. Πρώτοι και για αυτούς που εκτοπίζονται μέσα στην ίδια του τη χώρα. Πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες, παιδιά, ασυνόδευτα. και είδαμε πώς γίνεται η κατανομή τους σε φτωχές χώρες. Άρα υπάρχει αυξημένη ανάγκη για παιδεία έτσι. Και φυσικά το τελευταίο που χρειάζεται είναι να έχουμε τις τετριμένες στατικές, τα ίδια για τα ίδια, μήπως καλύψουμε αυτούς τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο επίσης για το σύστημα το εκπαιδευτικό. Γιατί εδώ πέρα μπαίνει το ποιοτικό στοιχείο. Σε κάποιες χώρες δεν είναι υποχρεωτική η παιδεία. Σε κάποιες χώρες πάνε στο δημοτικό τα παιδιά πολύ αργότερα από ό,τι στην Ευρώπη. 15-16, επομένως αυτοί οι άνθρωποι στερούνται παιδείας. Να, το ερώτημα είναι γιατί δεν έχει σημειωθεί πρόοδος και γιατί υπάρχει κενό στη χρηματοδότηση. Εδώ και χρόνια διαπιστώσαμε ότι έχουμε 39 δις κενό χρηματοδότησης κάθε χρόνο. Οπότε θα πρέπει οι δωρητές να εξαπλασιάσουν τη συμβολή τους για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα όσα έχουν ε, υποσχεθεί και να πετύχουμε τους σχετικούς στόχους. Είπαμε τι είχαμε με αυτούς τους στόχους, το 4% του ΕΒ για την παιδεία, το 15% του συνόλου των δαπανών για την παιδεία. Διαπιστώνεται ότι πάρα πολύ λίγες χώρες πέτυχαν να φτάσουν αυτούς τους στόχους ή κριτήρια. Και αυτό να δείχνει και από μια πρόσφατη άλλη μελέτη μας σε κάποια διάσκεψη που έγινε πάλι στον Τεκάρ. Λόγω και περισσότερο εστιαζόμαστε σε χρηματοδότηση επί τη βάση των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι σημαντικό. γιατί οι έρευνες κατέδειξαν ότι αυτό μπορεί να φέρει πάρα πολλές μαθήμετες συνέπειε. για τους πιο ευάλωτου, του πιο τέλο πάντων μη προνομιούχους, για αυτούς που είναι ανήμποροι μπροστά στο πρόβλημα. Είπαμε, αύξηση, όχι, μείωση διορθώνει, του μεγέθους των τάξεων του σχολείου. Και αυτό για να γίνει θέλει κατάλληλε υποδομές. Χρειάζεται επέμβαση λοιπόν, με αυτή την έννοια. Και τον εστιαζόμαστε στα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει από το να προσέχουμε και τα, τις ποιοτικές επιδόσεις. Πρόβλημα επομένως το πόσο εισφέρουν τα νοικοκυριά, το πρόβλημα είναι και το δημογραφικό, όλα αυτά στην έκθεσή μας τα αναδεικνύουμε και είπαμε ότι κάτι το οποίο πραγματικά έχει σημασία είναι η υποχρέωση λογοδοσία δηλαδή να επισημαίνεται έτσι ποιο είναι το πρόβλημα και πώ μπορεί να διορθωθεί. Πώς θα βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα. Και προς τα εκεί κατευθύνουν τις προσπάθειές μας για να υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία και ο προσανατολισμός μας είναι το ποιοτικό, όχι το ποσοτικό θέμα. Χρειάζονται στοιχεία όμως που διέπονται από διαφάνεια, γιατί έτσι φαίνεται που πάσχει το σύστημα και που τα πάει καλά. Άρα έτσι αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας. Να επισημάνουμε που είναι τα προβλήματα, ε, τότε θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Just Πολύ σύντομα να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Πεγιό. Όντως, βάσισα την παρουσίασή μου σε ποσοτικά στοιχεία, σε αριθμούς για να δείξω πραγματικά ποια είναι η προσέγγιση των ΜΕΝ και των ΔΕ και είναι πολύ δύσκολο, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ε, να μπορέσει κανείς να βασιστεί με αποτελεσματικό και χρήσιμο τρόπο σε στοιχεία τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν γνωρίζουμε καλά. Όσον αφορά βεβαίως την ποιοτική προσέγγιση, έχετε δίκιο. Είναι πολύ σημαντική το κάθε σύστημα το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα έχει το δικό του τρόπο αξιολόγησης, τις δικές του παραμέτρου και κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει με ένα ομοιογενές σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες όλων αυτών των συστημάτων, να δούμε ποια είναι τα κριτήρια, ποιοι είναι οι δείκτες. Δεν μπορούμε να έχουμε μία στάνταρ προσέγγιση που τα ε, αξιολογεί με τον ίδιο τρόπο όλα τα συστήματα. Την κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση. Παραδείγματο χάρη, το θέμα των φύλων. Μιλήσαμε για τον Ήγηρα, μιλήσαμε για την ενσωμάτωση, παραδείγματο χάρη στα νέα προγράμματα των ε, κοριτσιών και πώς ε, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαιτερότητες, ε, τα εμπόδια και τα προβλήματα της κάθε χώρας. Σας έδωσα εξάλλου λίγα παραδείγματα γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί εμείς ήμασταν οι πρώτοι που ανακοινώσαμε το ποσό που θα διαθέσουμε. Το υποσχεθήκαμε και το δεσμεύσαμε και στείλαμε ένα πολύ ε, σοβαρό αν θέλετε μήνυμα σε όλους τους συγχρηματοδότες, τους συναδέλφους, στους εταίρους μας και είμαστε πολύ ψηλά στον κατάλογο των ε, δωρητών, των ε, χρηματοδοτών στον τομέα της υγείας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα τρία δις φέτος. Αλλά είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος μεν, ελπίζουμε να τον ε, φτάσουμε. Από την άλλη εννοείται ότι δεν αρκεί το ποσό αυτό για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται πολυμορφία και υπάρχει πολυμορφία των δωρητών, αυτών που συνεισφέρουν με διαφορετικούς τρόπους, σε διαφορετικά επίπεδα, στην στήριξη των προσπαθειών για ενίσχυση της εκπαίδευσης. Εκατομμύρια από κάθε είδους νόμισμα συγκεντρώνονται. Προσπάθειά μας είναι ταυτόχρονα να ενσωματώσουμε και την τεχνική βοήθεια και την εμπειρογνωμοσύνη ε, καλύτερη πρόσβαση για τις πιο ευάλωτες ομάδες, να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για όλες αυτές τις περιοχές που πλήττονται ακόμα από κρίση, από συγκρούσεις. Προσπαθούμε δηλαδή να πολλαπλασιάσουμε τις πρωτοβουλίες, τις ε, προσπάθειες και τους τρόπους συνεισφοράς. Για πρώτη φορά ξεκινήσαμε έναν καινούριο διάλογο μεταξύ αυτών που συνεισφέρουν σε αυτές τις προσπάθειες μέσω της πλατφόρμας που σας παρουσίασα αλλά και άλλων παρόμοιων τεχνικών, δυνατοτήτων όπως αυτή η πλατφόρμα. Αυτό βοηθάει πολύ. Συζητούμε, συμβουλευόμαστε, και βεβαίως και μέσω της διμερούς στήριξης, συγκεκριμένα με κάποιες χώρες, αλλά βεβαίως ε, συνεργαζόμαστε και μέσω των ε, αντιπροσωπιών μας, των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου στις χώρες τις οποίες στηρίζουμε και προσπαθούμε κάθε φορά να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας με άλλες ε, διεθνείς ε, πρωτοβουλίες. Παραδείγματο χάρη στην Ζιμπάμπουε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει και συντονίζει γενικότερες προσπάθειες οι οποίες ξεκίνησαν από άλλες πηγές. Λιγότερο από το 2% της ανθρωπιστικής βοήθειας καταλήγει σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτά είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε. Μπορώ να τα ελέγξω και να σας πω αν συνεχίζουν να είναι αυτά. Εννοείται βεβαίως ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Πριν από δύο χρόνια το ποσό αυτό ήταν 15 με 20 εκατομμύρια. Έχει φτάσει τα 100 και προσπαθούμε να αυξήσουμε το ποσό αυτό και βεβαίως να δεσμεύσουμε τα ποσά έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο ε, που πραγματικά θα βοηθήσει. Ο κύριος Γκέρενς ρώτησε για την αναπαραγωγική υγεία, μίλησε για τα σεξουαλικά δικαιώματα, τη στήριξη των ε, νέων κοριτσιών για όλα τα θέματα αυτά που αφορούν την σεξουαλική τους υγεία, τη δυνατότητα που πρέπει να τους δίνεται να αποφασίσουν, να προστατευθούν. Χρειάζεται υποδομή, βεβαίως χρειάζονται ιατρία, νοσοκομεία, ιδιαίτερα για περιοχές ε, στην Αφρική, στην Ήπεθρο, ιδιαίτερα για την κάλυψη των αναγκών στις νέες μητέρες πριν τον τοκετό. Κυρία Μακάβριν. Η απάντησή μου είναι ότι βεβαίως έχουμε δικά μας ε, προγράμματα, ότι χρηματοδοτούμε και άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και προσπαθούμε να αναπτύξουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούν τον τομέα της υγείας. Παραδείγματος χάρη θέματα που αφορούν τα σχολικά γεύματα, τις καντίνες, το πώς ε, οι οικογένειες με παιδιά, με πολλά παιδιά, οι οικογένειες ε, με συγκεκριμένες ε, και περιορισμένες δυνατότητες να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Προσφέρουμε ειδικά προγράμματα για την καθαριότητα. Και βεβαίως εδώ ο ρόλος ε, των ε, φορέων του ιδιωτικού τομέα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ξέρετε ότι το πιο σημαντικό, αν θέλετε, που θα πρέπει καταρχήν να ξεπεράσουμε είναι το ρεφλέξ που έχουν ακόμα πολλές οικογένειες, ιδιαίτερα πολίτεχνες οικογένειες να στέλνουν μόνο τα αγόρια στο σχολείο και όχι τα κορίτσια, καθότι η εκπαίδευση συνεχίζει να αποτελεί ένα βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με ποιο τρόπο λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια, τις δυσκολίες, να βελτιώσουμε την πρόσβαση των οικογενειών στα σχολεία. Καταρχήν ξεκινώντας έναν διάλογο μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης, των δωρητών, για να αποφύγουμε επικαλύψεις. Βεβαίως, εμείς είναι δύσκολο να χρηματοδοτήσουμε μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις χώρες χωρίς προηγουμένως να υπάρχει απόφαση αυτών των χωρών, των εθνικών αρχών. Γι' αυτό και προσπαθούμε να συνεργαστούμε εκ των προτέρων με τις αρχές ε, των χωρών αυτών, τα Υπουργεία Παιδείας και τις αρμόδιες επιτροπές. Ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσεις σας. Έχετε ακόμα ένα λεπτό. Ένα τελευταίο σχόλιο. Γιατί πρέπει να το πω. Με ρωτήσατε τι κάνουμε που να αλλάζει την κατάσταση. Νομίζω ότι η ερμηνεία της εκπαίδευσης ε, ως δημόσιο αγαθό και όχι ως ιδιωτικό αγαθό. Δηλαδή προσπαθήσαμε να υπάρχει μια δαπάνη για την εκπαίδευση ε, η οποία θα συνδέεται με την ανάπτυξη ε, και όπως είπα είναι ε, δημόσιο και όχι ιδιωτικό αγαθό. Αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερο, ε, να κάνουμε ακόμη περισσότερο, ήταν να χρησιμοποιείται η δαπάνη για την εκπαίδευση όπου χρειάζεται περισσότερο, στις στοχότερες χώρες και όταν μπορεί η επέμβαση αυτή πραγματικά να βοηθήσει τις χώρες να βγουν από το περιθώριο στο οποίο βρίσκονται το πώς θα το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε αυτό σημαίνει ότι βελτιώνουμε και την ε, αίσθηση κυριότητας που έχουν αυτές οι χώρες ε, του συστήματος εκπαίδευσής τους. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο επόμενο πάνελ της συζήτησή μας, του οποίου συντονιστής ε, θα είναι ο Βανσόν Πεγιόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρώτο αυτό πάνελ και την πρώτη αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε πόσο πολλά είναι τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Ε, στο δεύτερο αυτό τμήμα, στο δεύτερο πάνελ της συζήτησής μας, έχουμε τρεις ε, προσκεκλημένες. Θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Μήπως παρακαλώ μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτησή σας ε, εκτός αίθουσας. Ευχαριστώ. Αλεξάνδρα Μακάροφ είναι η πρώτη προσκεκλημένη μας ε, που δουλεύει στη UNICEF και ειδικότερα στις σχέσεις με τους ε, ε, θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακούσουμε λίγο περισσότερα για το θέμα αυτό ή για τα διδάγματα που μπορούμε να λάβουμε από τις επιτόπου εμπειρίες. Κάρικ Βίτιγκ, η οποία είναι ε, οικονομολόγος ε, και τμήματάρχης ε, της γερμανικής επιχείρησης διεθνούς συνεργασίας που θα μας μιλήσει για την αναθεώρηση της αγοράς εργασίας και έχουμε επίσης και μία τρίτη προσκεκλημένη, την Ινές Τζεμάλη από την Plan International η οποία δεν ασχολείται όμως μόνο με την εκπαίδευση αλλά ε, ασχολείται κυρίως με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των νέων γυναικών. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό επειδή όλο και περισσότερο το βλέπουμε στις στατιστικές. Δεν μας κάνει εντύπωση ειδικότερα σε υποανάπτυξη χώρες αλλά και στις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι οι νέες γυναίκες υποφέρουν ιδιαίτερως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα μας μιλήσει λοιπόν περισσότερο γι' αυτό. Η κυρία Μακάροφ θα αρχίσει και ε, μετά στο τέλος των τριών παρουσιάσεών σας ε, θα ακουστούν οι ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, την Επιτροπή σας που μας κάλεσε και προκειμένου να προσπαθήσουμε κι εμείς να άρουμε από κοινού κάποια εμπόδια της εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να συνεχίσω με κάτι θετικό. Ε, ενδεχομένως να θεωρούσα ότι θα είχε καλυφθεί ενδεχομένως από το προηγούμενο πάνελ, αλλά μάλλον ε, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Ε, ίσως αυτό όμως θα μπορέσει να ε, ε σας δώσει και κάποια επιχειρήματα όταν κάποιοι, μιλάτε με κάποιους που είναι λιγότερο πεπισμένοι ως προς τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση. Θα αρχίσω λοιπόν με ένα πολύ απλό πράγμα. Ένα δισεκατομμύριο ε, ένα, ένα δισεκατομμύριο άτομα τα οποία δεν συμμετέχουν στη σχολική εκπαίδευση φέτο. Ένα δισεκατομμύριο λόγοι λοιπόν να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Κάτι ακόμη είναι ανθρώπινο δικαίωμα η εκπαίδευση. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να πάει σχολείο. Ε, γιατί δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να βγουν από τη φτώχεια και τους υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον. Όμως το να το συνδέσουμε αυτό με την ανάπτυξη είναι κάτι το λογικό, αλλά είναι και ο καλύτερος τρόπος ε, για την ε, ε, χειραφέτηση του καθενός, γιατί ένα κάθε έτος εκπαίδευσης δίνει 10% αύξηση στην, στα, στα έσοδα του κάθε ανθρώπου. Συνεπώς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αφορά όμως μόνο την οικονομική, το οικονομικό αποτέλεσμα η εκπαίδευση, αφορά το κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να μειώσει την θνησιμότητα των μητέρων, την ανισότητα μεταξύ των φίλων και πολλά ε, άλλα ε, να αντιμετωπίσει πολλά άλλα προβλήματα που ε, υπάρχουν σήμερα. Είναι ένας τρόπος βελτίωσης της κατάστασης για τις μελλοντικέ γενναίες και είναι ένας καλύτερος τρόπος ε, ένταξης του ατόμου αλλά και των οικογενειών του στην κοινότητα στην οποία ανήκουν. Το να υπάρχει λοιπόν υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης σε όλους, σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια υπό το στόχο 4 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικότερα ε, στη σημερινή ε, συγκυρία όπου τα οικονομικά, οικονομικές δυσκολίες μπορεί να μειώσουν τα χρηματοδοτικά μας μέσα ε, και ειδικότερα επειδή επηρεάζεται η εφαρμογή των προγραμμάτων που θα οδηγούσαν στην επίτευξη του στόχου 4. Πρόθεση λοιπόν της οικουμενικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες Εκτός λοιπόν από το κοινωνικό κομμάτι ε, υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα, πολλά εμπόδια που την παρεμποδίζουν. Μπορεί κάποιος να πει και την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση ότι να λέμε ότι ο μόνος λόγος είναι η μικρή χρηματοδότηση. Είναι όμως ε, και άλλοι λόγοι, όπως η κακή ποιότητα της εκπαίδευσης. Δεν θα μπορέσω να τους καλύψω όλους σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τους καλύψει όλους σε μία ομιλία, γιατί είναι τόσοι πολλοί. Θα αναφερθώ όμως στις δημογραφικές τάσεις και στην ανισότητα που υπάρχει. Η δημογραφική ανάπτυξη είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη πρόκληση που είναι μερικές φορές πιο σημαντική από την ίδια την εκπαίδευση γιατί το γεγονός ότι ε, αυξάνονται δημογραφικά κάποιες χώρες δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Στην υποσαχάρια Αφρική θα πρέπει 450 εκατομμύρια παιδιά ε, από έως 15 ετών να πάνε στο σχολείο μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα έπρεπε να υπάρξει και μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ε, κάτι το οποίο η χώρα δεν ε, έχει πάντοτε ούτε τα μέσα ούτε τη θέληση να το κάνει. Όσον αφορά το επίπεδο εκμάθησης, είναι πολύ χαμηλό σε πολλές χώρες, ειδικότερα σε χώρες χαμηλού εισοδήματος ε, και η αδυναμία της συμμετοχής στη μάθηση αρχίζει από πολύ νωρίς ένα ε, 90% ε, ε, ε, των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο. αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν τι απαραίτητε δεξιότητε για να μπορούν να είναι παραγωγικά στην ενήλικη ζωή του. Να έρθω τώρα στο κομμάτι τη ανισότητα, που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό για τη UNICEF και στο πλαίσιο του ότι κανένα δεν πρέπει να μένει πίσω. Ε, όσο φθηγότερη είναι η χώρα, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των ανισοτήτων. Τα παιδιά που αποκλείονται από την εκπαίδευση δεν προέρχονται από, από τι ίδιε κοινωνικέ ομάδε, συνήθω από τι φτωχότερε περιοχέ από τι περιοχέ τη υπαίθρου, είναι κορίτσια, ε, λόγω ε, της ε, εθνότητά του μπορεί να την χάνουν Ε, Υπάρχουν επίση προβλήματα αναπηρία που παρεμποδίζουν την, δυνα... την δυνατότητα των παιδιών αυτών να πάνε στο σχολείο. Είναι κάτι που συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικέ φορέ λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ανισότητα, όχι μόνο και όσον αφορά την χρηματοδότηση και το πώ κατανέμεται, αλλά και ως προς τις προτεραιότητες. Κάποιες χώρες ε, χαμηλού εισοδήματος ε, δίνουν περισσότερη χρηματοδότηση σε χώρες ε, που είναι ήδη κάπως, σε κάπως καλύτερη κατάσταση. Στο Μαλάου 68% των δημοσίων πόρων πηγαίνουν στο 10% των φοιτητών που σημαίνει ότι το 30% πρέπει να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο 90% των φοιτητών στο Μαλάου. Αλλά το να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση πιο περιθωριοποιημένα τμήματα του πληθυσμού δεν είναι επαρκέ για να λύσει το πρόβλημα. Πολλέ φορέ έχουν προκλήσει και στο ίδιο του το περιβάλλον όπω για παράδειγμα ασφάλεια, προβλήματα λόγω τη θρησκεία του. Ε, ε, πολλέ πολλές, οικογένειες πρέπει να κάνουν την επιλογή του κατά πόσο θα στείλουν τα παιδιά του να δουλέψουν ή θα τα στείλουν στο σχολείο, γιατί υπάρχει και το ζήτημα των εσόδων του νοικοκυριού, υπάρχει και το θέμα του ε, πρώιμου γάμου, γάμου σε πολύ μικρή ηλικία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με πιο ε, παραδοσιακά ε, ε, στοιχεία. το ίμιση των χωρών ε, που βγαίνουν από μια εμπόλεμη κατάσταση θα ξαναπέσουν σε μια κατάσταση εμπόλεμη σύγκρουση ε, εντός περίοδου 5 ετών, λένε οι έρευνες. Κάτι το οποίο λοιπόν πρέπει να ε, μας οδηγήσει στο να συμπεριλάβουμε και τον παράγοντα της ειρήνης στην όλη εξίσωση. η προσχολική εκπαίδευση. Αυτό είναι μια απαραίτητη αφετηρία για την αρχή της εκπαίδευσης και είναι και ένα πολύ καλό θεμέλιο για ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα, οπότε ενθαρρύνουμε την ΔΕΦΚΟ να επενδύσει στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά να έχει και μία προσέγγιση ε, κύκλου ε, ζωής. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες ε, στην προσχολική ηλικία, στις πρώτες τάξεις τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις επόμενες τάξεις και μετά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μία προσέγγιση κύκλου ζωής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις διάφορες ανάγκες των διαφόρων τμήματων του πληθυσμού. Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί και περισσότερη χρηματοδότηση ε, για την εκπαίδευση και σε μεθόδους που δίνουν περισσότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες εκμάθησης για, τους πιο, για τα πιο περιθωριοποιημένα παιδιά ε, για να μπορέσει η εκπαίδευση να αποδώσει όσον αφορά την ισότητα όλων των παιδιών, η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να κάνουν νέα κατανομή σημαντική σε μεγάλο βαθμό διαφορετική ε, των εκπαιδευτικών κονδυλίων και να υπάρξουν πολιτικέ που να είναι προσαρμοσμένε στην οικονομική κατάσταση τη χώρα. Να σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα από μια μελέτη τη UNICEF. Στι χώρε ε, χαμηλού εισοδήματο, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει τη σημαντικότερη επιρροή στην στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας για τις ΜΕΣΕΣ είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη της, την οικονομική της χώρας και για τις χώρες υψηλού εισοδήματος είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία έχει τη μεγαλύτερη επιρροή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τον τύπο τη επένδυση που πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε την ίδια, την ίδια επένδυση, την ίδια προσέγγιση για όλες τις χώρε ανεξαρτήτως εισοδήματο. Κάτι ακόμη πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι οι πολιτικέ υπέρ τη ισότητας <coughs> πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό το πρόγραμμα δεύτερη ευκαιρία, να δώσουμε δηλαδή στα παιδιά που είναι ε, αποκλεισμένα μία δεύτερη, εμπειρία, μια δεύτερη ευκαιρία, συγγνώμη, ε, επειδή υπάρχει και το χάσμα των γενεών και ίσως αυτό είναι ένας τρόπος να σταματήσει ο κύκλος της ε, ε, φτώχειας. Δεν χρειάζεται η φτώχεια να κληροδοτείται από γενιά σε γενιά δηλαδή οι ανάγκες ε, της πιο ε, ανεπτυγμένης, ας πούμε, του πιο ανεπτυγμένου τμήματος της νεολαίας ε, πρέπει να εξισορροπούνται με, τις, τα πιο φτωχά τμήματα του πληθυσμού και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται από τα πιο βασικά επίπεδα της εκπαίδευσης. Κάτι ακόμη, ενίσχυση των πρωτοβουλειών για την καλύτερη χρηματοδότηση, την αναθεώρηση του συστήματος ε, χρηματοδότησης της εκπαίδευση της χώρας, ειδικότερα στι χώρες που, που αρέχει βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης μια γεωγραφική ανακατανομή των ε, ε, πόρων. στο Μπαγκλαντέ, για παράδειγμα, έχουν εφαρμόσει μια πολιτική θετική διάκριση με περισσότερους δημόσιους πόρους αναφοιτητή σε φτωχότερε χώρε, κάτι το οποίο δείχνει ότι μπορούν ακόμη και σε μπορεί κανείς ακόμη και σε μια δύσκολη συγκυρία να επιτύχει το στόχο της ισότητας. Το να εγγράφονται περισσότερα παιδιά στο σχολείο σημαίνει ότι πρέπει να αρθούν κάποια εμπόδια, όπως για παράδειγμα το ότι πολλά παιδιά γίνονται γονείς, ε, παντρεύονται πολύ νωρί. Ε, πρέπει λοιπόν να γίνει μια κατανόηση της ε, κατάστασης των παιδιών αυτών και του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την κατανόηση χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες των παιδιών αυτών, κάτι που πρέπει να συμπεριληφθεί στα εθνικά συστήματα δεδομένων των χωρών. Να υπάρχει δηλαδή περισσότερο πληροφο... περισσότερη πληροφόρηση για τα παιδιά με αναπηρίες που είναι ένα μεγάλο κενό σε όλο τον κόσμο. Συμπερασματικά λοιπόν η άρση των εμποδίων, η ενίσχυση της πρόσβασης και οι καλές ευκαιρίες εκμάθησης όλα είναι απαραίτητα για να δοθούν στα παιδιά αυτό το ε, εκγενήσεως δικαίωμά τους που είναι η βασική εκπαίδευση. Merci euh, Σας ευχαριστούμε κυρία Μακάροφ. Λέει ο πρόεδρος. Και δίνει τον λόγο στην επόμενη ομιλία. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ την Επιτροπή Ανάπτυξης που μας κάλεσε. Λέω στην Γερμανική Υπηρεσία για την υλοποίηση της ε, τεχνικής αρρωγής στις όμορες ε, χώρες και εδώ και 40 χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται για την κατάρτιση και την παιδεία στον ε, αναπτυσσόμενο κόσμο. Πριν σας πω τις και τα προβλήματά μας, να σας πω πέντε μεγάλες επιτυχίες σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, το ΒΕΤ, αυτό που λέμε, <clears throat> παιδεία επαγγελματική κατάρτιση και μετά να σας αναλύσω ποιε είναι αυτέ οι, έξι προκλήσεις για τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλες χώρες. Και στο τέλος θα έχω κάποια σχόλια για γενικότερα προβλήματα στην αγορά εργασίας ε, σύμφωνα με την εμπειρία μας. Η πρώτη επιτυχία για αυτό το σύστημα ΒΕΤ αφορά την απασχολησιμότητα πολλών ανθρώπων στις αντισόμενες χώρες και όπως πάντοτε ισχύει, αυτό απαιτεί συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και θα πρέπει αυτό το σύστημα της κατάρτισης εκπαίδευσης να προσανατολίζεται προς την ε, ε, ζήτηση σε κοινέ αρμοδιότητες και ευθύνες. Επίσης χρειάζεται να υπάρχει ε, κατάρτιση και στο χώρο της εργασίας. Όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα στην απασχόληση σήμερα, οπότε χρειάζεται να αναπτύξει κανείς δεξιότητες απασχολησιμότητας. Άρα συνδυασμός ε, του κανείς στην πράξη να ξέρει τι γίνεται και να είναι και καταρτισμένος γενικότερα ούτως ώστε επαγγελματικά, μεθοδολογικά, κοινωνικά να είναι παρκής στο ότι απαιτείται. Άλλη επιτυχία, μπορεί να σας αναφέρω, είναι η αποδοχή από πλευράς της ε, κοινωνίας κάποιων προτύπων και χρειάζεται επίση μια εξέταση αυτών των προτύπων, ώστε να οδηγήσουν σε απόκτηση δεξιοτήτων. Πιστοποιήσεις, ό,τι βοηθάει για απασχολησιμότητα, κινητικότητα, κοινωνική αποδοχή. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην ισόβια κατάρτιση. Και έτσι να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά εργασίας. Τέταρτη επιτυχία. Εκπαιδευμένο προσωπικό, αυτή δηλαδή που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση. Και αυτοί που διδάσκουν στα σχολεία και στο χώρο εργασίας. Πέμπτον, να έχει θεσμικό χαρακτήρα η έρευνα και η, ο που παρέχεται. Να σας πω επομένως τι έχουμε διαπιστώσει από την εμπειρία μας σε σχέση με το τι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν στις αντισόμενες χώρες. Πρώτον, η δομή των επιχειρήσεων. Στις χώρες αυτές έχει πολλές μικροεπιχειρήσεις. Πολλές φορές όμως υπάρχει δισταγμός, υπάρχει ε, ε έλλειψη θέλησης για κατάρτιση. Όμως εμεί θα πρέπει να στραφούμε στις κοινότητες, να οργανωθούν και έτσι θα δούμε τι θα κάνουμε για τους οργανισμούς που δεν επενδύουν στην κατάρτιση. Τώρα να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το δουλευτικό σύστημα, έλλειψη συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και κράτους. Δύο τινά. Πρώτον, η εκπαίδευση από το σχολείο σημαίνει ότι το σύστημα θα είναι προσταλισμένο προς την ζήτηση. Όμως αυτό δεν αντιστοιχεί τώρα στην ποικιλία που υπάρχει ούτε στην ποικιλία των εταιριών, ούτε στη ζήτηση, ούτε σε εταιρείε. Οπότε υπάρχει κάποιο είδους παραπληροφόρηση μεταξύ ζήτησης και προσφοράς σε πολλές χώρες στις οποίες δουλεύουμε έχουμε κάποια προγράμματα που λειτουργούν με διαφορετική ορολογία. Οπότε άλλα ζητεί η δουλειά και άλλα δίνει η εκπαίδευση. Και έτσι διονύζεται μια τέτοια κατάσταση. τερίτη πρόκληση. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος ανεπαρκής κατάρτιση που οδηγάει σε εργασίες χαμηλού επίπεδου. Και έτσι τελικά η αυτού του είδους εκπαίδευση ε, αφορά μόνο αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα καλύτερο, αντί να τους καλύπτει όλους. Άρα χρειάζεται κατάρτιση στο σχολείο. Και χρειάζεται να συμπλέψουν για αυτές τις προσπάθειες οι εταιρείε και το σχολείο. Χρειάζονται περισσότερα κίνητρα. Πέμπτο πρόβλημα. Υπάρχουν ε, προβλήματα, υπάρχουν φραγμοί στο να πετύχει κανείς την ε, αλλαγή τη μετάβαση από την ε, βασική εκπαίδευση στην συνέχεια και στην κατάρτιση. Και μετά ε, από τις σχολές στη δουλειά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, κάποιος έχει δουλέψει, υπάρχουν άλλες ε, λήψεις στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και επίσης δεν υπάρχει προσανατολισμός, ε, οπότε χρειάζεται βελτίωση του συστήματος κατάρτισης, να εκμεταλλευτούμε τις επιτυχίες μας και έτσι να δούμε πώς θα έχουμε κάποιες δομές που θα προωθούν καλύτερα τους καταρτιζόμενους. Έκτη πρόκληση είναι οι υπερβολικές προσδοκίες, ότι δηλαδή το σύστημα της κατάρτισης μου λύσει όλα τα προβλήματα. ή τα συστήματα κατάρτισης είναι μόνο ένας από τους παράγοντες, μία από τις μεταβλητές. Επίσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολλές φορές δεν έχουν καλές επιδόσεις στην Αφρική. Ούτε αυτό μπορεί να το καλύψει μόνο η κατάρτιση και η εκπαίδευση. Μόνο την προσφορά εργασίας μπορεί να καλύψει. Δεν μπορούμε αυτό μόνο να θεωρήσουμε ότι βελτιώνοντας το ΒΕΤ θα έχουμε καλύτερε επιδόσεις στην απασχόληση. Τώρα θα δούμε κάποιου είδους γενικότερα προβλήματα για την αγορά εργασία να δούμε εμεί τι προτείνουμε για αυτά τα προβλήματα. Σε πολλέ από τις χώρε με τις οποίες εργαζόμαστε η ανεργία είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου των προβλήματων τη απασχόλησης. Άρα, μία από τις λύσεις θα ήταν να έχουμε κάποια προβλήματα, κάποια, συγγνώμη, κάποια προγράμματα κατά της εκπαίδευσης, ε, τα οποία να είναι κομμένα και μέσα στα μέτρα αυτών που είναι άνεργοι, να ταιριάζουν επίσης στις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη σε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι. Οπότε θα πρέπει κανείς να παρακολουθήσει ποια είναι τα προβλήματα στην ε, Ήπεθρο και πόσο εκεί δεν είχαμε καμία πρόοδο όσον αφορά τα έσοδα των οικοκυριών και την πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια. Άρα η απασχόληση μπορεί να βελτιωθεί εάν η ζήτηση και η προσφορά και οι ενεργές πολιτικές όλα μαζί ε, κατατείνουν στη λύση του προβλήματος. Άρα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της απασχόλησης. Να συνδυαστούν όλες αυτές οι μεταβλητές. Κατάρτιση, εκπαίδευση, να ληφθεί υπόψη αγορά απασχόληση, αλλά και το τι ζητάει ο ιδιωτικό τομέα. Άρα, να υπάρχουν καλές συνθήκες απασχόλησης και να βοηθήσουμε το πώς θα συντεριέξει καλύτερα η κατάρτιση της εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Και επίσης να οργανώσουμε καλύτερα ακόμα και το σύστημα των αιτήσεων απασχόληση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πραγματικά καταφέρατε με λίγο χρόνο ομιλίας να μας πείτε πάρα πολλά πράγματα. Μπράβο και θα δώσω το λόγο στην τελευταία ομιλήτρια. Good afternoon Καλό απόγευμα. σα ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο σήμερα. Ο σκοπό μα είναι πω θα χειραφετηθούν τα κορίτσια έτσι ώστε μέσα από την εκπαίδευση να βελτιωθεί η κατάσταση των κοριτσιών, η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταρχήν η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα 20 τελευταία χρόνια. Παραμένει όμως μεγάλη πρόκληση η ενσωμάτωση των κοριτσιών στην περαιτέρω εκπαίδευση δευτεροβάθμια και ανώτατη. Υπάρχουν ε, βεβαίως σημαντικές δυσκολίες και κρίσεις ε, στον τομέα της υγείας, στον τομέα της ανθρωπιστικής ε, κατάστασης και θα πρέπει καταρχήν να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα κορίτσια, εάν μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν τις ε, διανοητικές και σωματικές τους δυνατότητες, γιατί πολλές φορές υπολείπονται σε όλους αυτούς τους τομείς. Σημαντικό είναι καταρχήν να δούμε πώς θα δώσουμε θετικές εμπειρίες στα κορίτσια. Πώς ε, τα κορίτσια θα περάσουν από τη βασική πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην δευτεροβάθμια. Πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες σε κάποιες ε, κοινωνίες που θεωρούν ότι τα κορίτσια πρέπει να μένουν στο σπίτι. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν προκαταλήψεις και πολύ έντονες πιέσεις έτσι ώστε τα κορίτσια να μην μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση. Το σχολείο, βεβαίως, υπάρχουν πολλές φορές ε, επιπλέον προκαταλήψεις, διακρίσεις, κάτι που περιορίζει τα κορίτσια. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα νέα κορίτσια να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μετά τη βασική, την πρωτοβάθμια και βεβαίως να ενσωματωθούν στην αγορά της εργασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε θέσει σαν στόχο. Τα κορίτσια τα οποία μπορούν να ζήσουν με υγεία, με εκπαίδευση και με ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων τους, χειραφετημένα κορίτσια μπορούν να είναι στήριγμα ε, και βασική βοήθεια και για τις οικογένειές τους. Χρειάζεται καταρχήν να προσφέρουμε μία εκπαίδευση, μία παιδεία ποιοτική, η οποία να ενσωματώνει και τα κορίτσια. Εκπαίδευση η οποία να σέβεται τις σημαντικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει, όπως την ίση εκπροσώπηση αγοριών και κοριτσιών. Να μπορούν τα κορίτσια να έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αντιμετώπιση που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Θα αποκτήσουν δεξιότητες και προσόντα όπως ε, την ε, λήψη αποφάσεων, όπως τις ηγετικές ικανότητες και θα μπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειες και τις κοινωνίες τις οποίες ζουν. Τα κορίτσια θα πρέπει λοιπόν να περάσουν μέσα από μία εκπαίδευση, από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να προσφέρει ίσες δυνατότητες στα αγόρια και τα κορίτσια με εκπαιδευτικά συστήματα, με κατάρτιση και σεμινάρια εκπαιδευτικά στους δασκάλους, στους καθηγητές, που να εξαλείφουν και να καταπολεμούν τις φιλετικές διακρίσεις, τις σεξουαλικές διακρίσεις, τις διακρίσεις μεταξύ αγοριών και ε, κοριτσιών. Θεωρούμε ότι το κάθε κορίτσι θα πρέπει να μπορεί να μαθαίνει, να ενσωματώνεται σε μια κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης και να μπορεί κατόπιν να προγραμματίζει το μέλλον της, να ενσωματώνεται στην αγορά εργασίας. Και αυτό δεν μπορεί παρά να γίνει με την ενδυνάμωση των προσόντων, των δεξιοτήτων τους σε όλους τους τομείς και την αύξηση της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται ακόμα και σε περιοχές όπου επικρατεί κρίση η ίση εκπροσώπηση των αγοριών και των κοριτσιών δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την ίση αντιμετώπιση των κοριτσιών, των μικρών κοριτσιών από τα πρώτα χρόνια στο σχολείο. Θα πρέπει να αυξηθεί το τμήμα του προϋπολογισμού, των εθνικών προϋπολογισμών που διατίθεται στη βασική εκπαίδευση για την καλύτερη σωμάτιση των κοριτσιών. Γνωρίζουμε όμως ότι στις λιγότερο αναπτυγμένε χώρες, στις πιο φτωχές χώρες, δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός και τα κονδύλια για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα όπως οι διακρίσεις κατά των κοριτσιών. Προτείνουμε βεβαίως να στηρίξουμε αυτή τη χρηματοδότηση με διμερή χρηματοδότηση, με δωρητές οι οποίοι συγκεκριμένα θα χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα έτσι ώστε να ξεπεραστεί και να εξελιχθεί αυτή η διάκριση κατά των κοριτσιών με συγκεκριμένα προγράμματα, με προϋπολογισμούς που θα έχουν σαν στόχο να εξαλείψουν όλες αυτές τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, τους καταναγκαστικούς γάμους, την ε, υποχρέωση τα κορίτσια να παραμένουν στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλες αυτές οι διακρίσεις να πάψουν να υπάρχουν. Για μένα εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες μπορούν να ενσωματωθούν στη δευτερομάθημα και την ανώτατη εκπαίδευση και με αυτόν τον τρόπο να χειραφετηθούν και να στηρίξουν τις οικογένειες και την κοινωνία. Είναι σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι ο φεμινισμός, τα κινήματα για τη χειραφέτηση των γυναικών θα πρέπει εδώ να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Μία εκπαίδευση η οποία αλλάζει τη σχέση μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών είναι καθοριστική. Τα αγόρια και τα κορίτσια θα πρέπει να μαθαίνουν καλύτερα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο και εφόσον αντιμετωπίζονται με τις ιδιαιτερότητές τους. Η φωνή των κοριτσιών πρέπει να εισακουστεί. Η φωνή των κοριτσιών ε, μετράει, είναι σημαντική. Χρειάζεται να στηρίξουμε κάθε κίνημα που βοηθάει μικρά κορίτσια και τις ε, νέες κοπέλες να ενσωματωθούν καλύτερα με κάθε τρόπο στα προγράμματα κατάρτισης, στα προγράμματα ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας. Είναι καθοριστικό να ακούσουμε τα κορίτσια σε όλες τις φάσεις και τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμελήσουμε τα κορίτσια έτσι ώστε να μπορέσουν να μάθουν, να αποφασίσουν και να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Merci beaucoup pour euh, ces interventions. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, ομιλίες αυτές. Ε, για να συνεχίσω τον ε, προβληματισμό σας, Έχουμε συχνά άντρες οι δήμονες για θέματα οικονομικής ε, βοήθειας και χρηματοδότησης. Αυτή τη φορά είχαμε πέντε οι δήμονες γυναίκες. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε σήμερα, γιατί τα ε, επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση είναι γυναικεία επαγγέλματα και αυτό δημιουργεί στερεότυπα. Ε, και αυτό είναι δύσκολο. Για παράδειγμα, 90% των δασκάλων στο δημοτικό σχολείο στη χώρα μου είναι γυναίκες. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που ήταν πέντε εμπειρογνώμονες γυναίκες εδώ σήμερα. Αναρωτιέμαι παρόλα αυτά τι μπορεί να σημαίνει η απερίμωση του επαγγέλματος αυτού σε σχέση με τους άντρες, ότι οι άντρες δεν συμμετέχουν καθόλου αυτό το λέω για να συνεχίσω λιγάκι τον προβληματισμό σας. Να αρχίσουμε λοιπόν τώρα τη συζήτηση. Δεν, όποιοι συνάδελφοι θέλουν ε, να θέσουν ερωτήσεις ε, έχουν το λόγο. Κύριε Βεντά, ευχαριστώ. Το ερώτημά μου είναι προς την κυρία Βέντικ. ο ιδιωτικό τομέα και ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπός του είναι κάτι που το διαπιστώνουμε όλοι, αναφέρεστε πολύ συχνά σε αυτό και λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό ειδικότερα στον τομέα της ανάπτυξης. Πώς μπορούν οι επενδυτές, οι επιχειρήσεις να ενθαρρυνθούν να βλέπουν ε, την ευρύτερη εικόνα ε, και να ε, μπορούν να ε, προσαρμόσουν ε, τις, ε, τα διάφορα project που εφαρμόζουν τους στόχους για να βελτιώσουν την κατάσταση του πληθυσμού των χωρών αυτών. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποια ανάγκη και για τέτοιου είδους εκπαίδευση, μια τέτοιου είδους παιδαγωγική ανάγκη γιατί έχει να κάνει νομίζω και με το θέμα των προσόντων, των επαγγελματικών προσόντων των διδασκάλων και επίσης τι ε, μπορεί να γίνει ώστε να ε, αποφευχθεί η έλλειψη διδασκάλων. Η κυρία Μακάβαν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσαμε πάρα πολύ για τα σχολεία στο πρώτο πάνελ ε, του, της σημερινής συνεδρίασης. Ε, αν σκεφτεί κανείς τη σύνοδο του Αμπιτζάν, ε, το θέμα ήταν πώς οι νέοι άνθρωποι θα συμμετέχουν καλύτερα στην αγορά εργασίας, ε, στην Αφρική. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ είναι εδώ ακόμη, θα μπορούσε να μας πει λίγο περισσότερο πώς θεωρεί ότι αυτό το θεματολόγιο θα προχωρήσει όλο αυτό το θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους ανθρώπους, όχι μόνο για το θέμα της σχολικής εκπαίδευση και για τα projects. Νομίζω ότι επειδή μόλις γυρίσαμε από την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ε, είδαμε ένα-δυο παραδείγματα μικρών τοπικών projects από ντόπιου πληθυσμού και όχι από μεγάλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είδαμε πάρα πολύ ε, καλούς και έξυπνους επιχειρηματίες νέοι. νέοι. ένας ας πούμε είχε εφεύρει μία μηχανή που ξεφλούδιζε τα φιστίκια και ρωτήσαμε εκεί τους τοπικούς υπευθύνους ε, αν μπορούμε κάπως να ενισχύσουμε αυτήν την ε, ε, καινοτομία των ανθρώπων αυτών. Ήταν πάντοτε πάρα πολύ περίπλοκο γιατί υπήρχαν πάρα πολλές απαιτήσει όσον αφορά τα προγράμματα, πρέπει να περνάμε μέσα από μεγάλους οργανισμούς. Δεν έχουμε δηλαδή καμία διευκόλυνση ενίσχυσης των ανθρώπων αυτών επιτόπου σε κάτι που κάνουν στη χώρα τους το ίδιο πρόβλημα το είχαμε και στην περιφερειακή πολιτική στο παρελθόν ε, όταν, ε, όταν ε, συζητούσαμε για την οικονομική αναδιάρθρωση. Πάντοτε τα χρήματα πήγαιναν σε μεγάλους οργανισμούς που είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των τοπικών αναγκών γιατί ήταν πάρα πολύ μακριά από αυτές τις τοπικές κοινωνίες. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και ε, ξέρω ότι ένα από τα προβλήματα του λογιστικού ελέγχου είναι ότι είναι πάντοτε στους τίτλους των εφημερίδων. Αν όμως θέλουμε ε, να ε, γίνει κάτι επιτόπου πρέπει να ανταποκρινόμαστε άμεσα. Και έχω ακούσει επίσης ότι είναι περισσότερο δαπανηρό κιόλα το να βοηθήσει κανείς κάποιον επιτόπου περνώντας από έναν τεράστιο ε, ε, οργανισμό που βρίσκεται τόσο μακριά. Γιατί πρέπει να περάσουμε πρώτα από τους διεθνείς μη κυβερνητικού οργανισμούς μέχρι να φτάσουμε στο τοπικό επίπεδο, από πάνω προς τα κάτω δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Βέντιξ σε σχέση με τέτοιου είδους projects. Βρίσκεται, βλέπετε τέτοιου είδους παραδείγματα άμεσης ενίσχυσης ε, ντόπιων κάποιων επιχειρηματιών. Όταν είχαμε πάει στην Κένια, για παράδειγμα, οι νέοι άνθρωποι ε, σε κάποιους ε, καταβλισμούς ε, έχτιζαν τουαλέτες και ντους για να μπορεί ο κόσμος να πλένεται. Είναι ένα, και αυτό ένα πολύ μικρό project. Αν σκεφτεί κανείς δηλαδή την πραγματικότητα το, της ζωής σε πολλές από αυτές τις κοινότητες, το να μπορεί κανείς ας πούμε να έχει μια πολύ πολύ μικρή επιχείρηση είναι ενδεχομένως το καλύτερο για ε, τον κόσμο εκεί. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε σε αυτούς τους όρους και θα ήθελα να μου πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει σχεδιάσει ε, ως συνέχεια στο Αμπιτζάν ώστε να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ωραία. Ποιος, ε, ποια θέλει να αρχίσει. Κυρία Βέντιχ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, βλέπω την άμεση ανίσχυση στις τοπικές ε, επιχειρήσεις ε, σε πολλά projects ε, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας. Όμως θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιτυχία όλου αυτού του εγχειρήματος. Προφανώς υπάρχουν ποικίλε προσεγγίσεις ε, πολύ, ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ε, όμως βάσει όλων αυτό που έχουμε δει κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι, είναι πολύ επιτυχή όσον αφορά ε, όσον αφορά την ανάπτυξη, την, την έναρξη των επιχειριών, αλλά μετά δεν συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις πολύ από την, ε, πολύ παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα <coughs> έχει επικεντρωθεί σε αυτό ακριβώς το στοιχείο. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ανέφερα κατά το τέλος της πολύ σύντομης παρουσίασής μου προσπαθεί να καλύψει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να ενσωματώνεται οποιαδήποτε τεχνική αρρωγή και επιστημονική βοήθεια στην ε, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ε, άτυπη ή επίσημη, και μάλιστα ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, να εξασφαλίσουμε ότι η υποστήριξη δεν είναι κάτι που συμβαίνει άπαξ. Μια άπαξ επέμβαση είτε προς την πλευρά της προσφοράς είτε προς την πλευρά της ζήτησης και η προσφορά και η ζήτηση πρέπει κάπως ε, να ε, αξιολογούνται σε σύγκριση μία με την άλλη ε, και σε εθνικό επίπεδο και σε σχέση με την έβρεση εργασίας ε, αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα ήθελα να το τονίσω. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχει κάποια συνέχεια στην, ε, στις υπηρεσίες της υποστήριξης που παρέχουμε μέσω της προώθησης πλατφορμών και κόμβων επιχειρηματικών που ελπίζουμε ότι θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και μετά από την ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου. Είτε με τα επιμελητήρια συνεργαζόμαστε, είτε με μικρές με, ε, οργανώσεις επιχειρήσεων στο πλαίσιο πάντοτε της ε, επαγγελματικής κατάρτισης και των σχετικών προγραμμάτων. Για να συμπληρώσετε την απάντησή σας, θα ήθελα να σας κάνω και εγώ μία ερώτηση. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Εντάξει, η κατάρτιση είναι σήμερα μία αγορά, υπάρχει μία ανάπτυξη τρομερή της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εις βάρος των δημοσίων επενδύσεων, γιατί ε, τα παιδιά των πλουσιότερων μπορούν να συμμετέχουν σε σπουδές που είναι επιπληρωμή. Ε, και εμείς ε, με τις μεγάλες μας και σημαντικές μας ε, σχολές βλέπουμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη λογική και στις χώρες του Μαγκρέμπ αλλά και στην Υποσαχάρη Αφρική για τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια. Κάτι κρύβεται πίσω από αυτό και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Στις αγορές τη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευσης ε, αντιμετωπίζετε συχνά μερικά ερωτήματα αρκετά δυσάρεστα που έχουν να κάνουν ε, με τη διαφθορά Αυτή τη στιγμή λοιπόν μία σχολή γίνεται μία τεράστια αγορά και το ξέρουμε αυτό στην Αφρική υπάρχει και είμαστε πλέον σε ανταγωνισμό και με τους Κινέζους φίλους μας και με τους Ιάπωνες φίλους μας που μόλις επένδυσαν πάρα πολλά ε, στην ε, Αίγυπτο αλλά και μεταξύ μας οι Γάλλοι με τους Γερμανούς κλπ. Εγώ επειδή ήμουν, προ... Ε, ήμουν υπουργό, είχα δει αυτόν τον ανταγωνισμό τον είχα ζήσει στο πετσί μου. Λοιπόν, μιλάμε ότι 15-20 δις ε, ε, ευρώ δεν ήταν επαρκή για να μας ε, καλύψουν και να μπορέσουν να μας λύσουν το πρόβλημα. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε, γιατί εδώ και δύο-τρία χρόνια εγώ νιώθω ότι όλο και περισσότερο οικονομικοί φορείς ε, πηγαίνουν στο, στην αγορά της εκπαίδευσης για να κερδίσουν χρήματα και είναι κάτι το σημαντικό και το λέω αυτό σε σχέση με αυτό που είπε ε, ο συνάδελφος προηγουμένως ε, μήπως έχει αυτό να κάνει με το όλο ζήτημα των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Και δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση με την ερώτησή μου αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή εγώ προέρχομαι από το εκπαιδευτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρω τι εννοείτε. Όχι, όχι, όχι, δεν με φέρνετε καθόλου σε δύσκολη θέση με την ερώτησή σας. Ε, η προώθηση ενός διτού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Αυτό θέλω να το τονίσω. Εμεί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στον οργανισμό μα με τι χώρε εταίρου μα είναι καλύτερη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά τεράστια συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλλά δεν σημαίνει ούτε και τεράστιες επιδοτήσεις από το δημόσιο τομέα. Η ισορροπία λοιπόν εξαρτάται, μεταξύ των δύο εξαρτάται από την ε, οικονομία, από το επίπεδο οργάνωσης ε, των ε, εργοδοτών και των επιχειρήσεων και από την ποιότητα του σχολικού συστήματος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ώρα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μεγαλύτερη όμως συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αντιβαίνει στην ανάπτυξη ορισμένων από τις τάσεις που αναφέρατε, γιατί ε, συμβαδίζει με την κατανομή των ευθυνών, την συγκέντρωση πόρων και την ανάπτυξη μιας κοινή γλώσσας μεταξύ των ε, επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού τομέα και αν αυτό είναι ενσωματωμένο στις αρχές ε, της κατευθυντήριες μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση και ενδεχομένως να παρεμποδίσει την ανάπτυξη των τάσεων που αναφέρεται. δεν το βρίσκω τεράστιο πρόβλημα για την ώρα. Ευχαριστώ. Maybe just, um, quickly to come back on the... Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι αποφάσισα να μιλήσω περισσότερο για τα πρώτα χρόνια στο σχολείο γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στο πώς περνούν τα νέα αγορία και κορίτσια από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας. Αλλά μιλώντας γι' αυτό, ξεχνάμε τα πρώτα χρόνια των παιδιών στο σχολείο. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό με την μεσοπρόθεσμη αυτή ακτίμηση, αξιολόγηση που κάνουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πρώτα χρόνια είναι καθαριστικά. Αν δεν ξεκίνησε η ενσωμάτωση σε ένα σχολείο των παιδιών πολύ νωρίς, έχουν σίγουρα καθυστερήσει και χάσει σημαντικές ευκαιρίες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να το συνειδητοποιήσουμε πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση για την επαγγελματική κατάρτιση. Ευχαριστώ πολύ με όλα αυτά που είπε η κυρία Μακέβαν. Πιστεύω ότι αυτές οι τάσεις πρέπει να στηριχθούν, να αξιολογηθούν από μας. Είναι πολύ σημαντικό στα πρώτα χρόνια της ενσωμάτωσης των παιδιών στα σχολεία να στηρίξουμε ιδιαίτερα την ενσωμάτωση περισσότερων κοριτσιών. Τα κορίτσια είναι μια ευάλωτη ομάδα. Πολλές φορές το ξεχνάμε. Χρειάζονται λοιπόν ιδιαίτερα προγράμματα, ιδιαίτερα για τις κοινωνίες αυτές που δεν θεωρούν ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών είναι προτεραιότητα. you. So, uh, you asked how, how companies can be... Thank you. Κάρατε και μια άλλη ερώτηση. Πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να δεσμευθούν. Καταρχήν σε ένα σύστημα που λειτουργεί με εκπαιδευτικό σύστημα και επαγγελματική κατάρτιση, Βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις ε, ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας εργασίας, αναπτύσσοντας και προσαρμόζοντας τα εκπαιδευτικά συστήματα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες αγοράς. Γιατί δεν λειτουργεί σαν αυτός σκοπός και απομονωμένο το Υπουργείο Παιδείας μιας χώρας, κοιτάει πάντα τι χρειάζεται η αγορά, τι ζητάει η αγορά για να προσαρμοστεί. Σίγουρα λοιπόν μονίμως χρειάζεται μια επαγγελματική κατάρτιση η οποία να βοηθάει όλους τους εργαζόμενους, τους νέους εργαζόμενους αλλά και όλους τους εργαζόμενους να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς εργασίας. Εννοείται ότι αυτό έχει ένα κόστος και οι επιχειρήσεις πρέπει να υπομισθούν ένα τμήμα αυτού του κόστους. Βεβαίως υπάρχουν ε, τα αποτελέσματα της κατανομής της παραγωγικής εργασίας, ο δημόσιος τομέας, ο οποίος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στην επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και το ρόλο των ε, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. χρειαζόμαστε καθηγητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές οι οποίοι να μπορούν να πάνε στις επιχειρήσεις και να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων και των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρουν αυτοί οι καθηγητές, αυτοί οι εκπαιδευτικοί και χρειάζεται μια πραγματική μεταρρύθμιση έτσι ώστε να ενσωματώνονται γρήγορα και με σωστό τρόπο τα μηνύματα που στέλνει η αγορά εργασίας. Και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειάζονται σωστά καταρτισμένοι ε, εκπαιδευτικοί. Όσον αφορά τις προκλήσεις, πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχει μια προθυμία από μέρους ε, των επιχειρήσεων ε, ιδιαίτερα όταν τους ζητούμε να επενδύσουν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Και αυτό που τους λέμε πάντα είναι ότι αυτό που κάνετε είναι άδικο και είναι και εγωιστικό, διότι προσπαθείτε να προσελκύσετε στις εταιρείες σας άτομα με προσόντα, με δεξιότητες, στους οποίους δεν έχετε συνεισφέρει καθόλου όσον αφορά την απόκτηση αυτών των προσόντων. Και νομίζω ότι έχουμε επιχειρήματα για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές να συνεισφέρουν. Κάτι που δεν ακούσαμε είναι πώς μπορούν οι ίδιοι οι νέοι να συμμετέχουν. Ήμουν πριν από λίγα χρόνια στο Τιμόρ, στην Ήπεθρο. Και προσπαθήσαμε να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν, πώς μπορούμε να προσελκύσουμε νέους στις αγροτικές εργασίες με ένα πιο τεχνολογικά προηγμένο τρόπο διαπιστώσαμε ότι σίγουρα χρειάζονται και άλλες δραστηριότητες όμως, όχι μόνο η γεωργία, όχι μόνο ο αγροτικός τομέας, το μάρκετινγκ, η πρόθεση των προϊόντων του στην αγορά κτλ. κτλ. Και αυτό βεβαίως το ανακαλύψαμε ακούγοντας τους ίδιους τους νέους, οι οποίοι ήθελαν να ενσωματωθούν σε άλλους τομείς της οικονομίας και να ε, αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες και προσόντα. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι να προσφέρουμε κάτι στους νέους, αλλά να ακούμε και τα δικά τους αιτήματα. Τελικά αυτό ήταν και η ερώτησή μου. Ο ιδιωτικός τομέας, ο καθαρά ιδιωτικός τομέας σε χώρες όπως η Αφρική, μπορεί να κινητοποιηθεί. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι ένας τεράστιο, ένα τεράστιο τμήμα της οικονομίας αυτών των χωρών εξαρτάται από τη γεωργία. Από την διατροφή, τα είδη διατροφής, την παραγωγή τους και την διανομή τους και διάθεσή τους στην αγορά. Και βλέπουμε ότι ο τρόπος πρόθεσης αυτών των προϊόντων διανέμοντάς τα παραδείγματο χάρη και σε άλλες ε, γειτονικές αγορές, δημιουργώντας νέα κανάλια πρόθεσης. Σίγουρα δεν είναι καθαρά γεωργικές, αν θέλετε, δραστηριότητες, αλλά σίγουρα συνδέονται και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την γεωργική παραγωγή. Πώς λοιπόν ε, μπορείτε να ενσωματώσετε τις αγροτικές αυτές δραστηριότητες, την αγροτική οικονομία, σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας των αφρικανικών χωρών, παραδείγματο χάρη. Και πώς μπορούμε να προσφέρουμε σεμινάρια επαγγελματικά κατάρτισης που να είναι κοντά μεν ε, στην αγροτική παραγωγή, στη γεωργία, αλλά διαφορετική τομείς οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με αυτόν τον πρωταρχικό, αν θέλετε, τομέα της παραγωγής τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι και οι πέντε ομιλητές ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Και εγώ ολοκληρώνοντας θα πω ότι σε καμία περίπτωση δεν καλούμεθα εδώ να επιλέξουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκπαίδευσης. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όλο το περιβάλλον, τους τομείς όπως ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, οι μεταφορές. Και βεβαίως η δυνατότητα επιλογών Υπάρχουν χώρες σήμερα, στη Βόρεια Αφρική παραδείγματος χάρη, που έχουν πολλούς νέους πτυχιούχους, άνεργους. Είναι μια τραγική κατάσταση. Και όλα αυτά δεν πρέπει να τα αγνοούμε στα μοντέλα που προτείνουμε. Στόχος μας είναι τα ποσά που δαπανούνται τα οποία μπορεί να μην έχουν αυξηθεί, αλλά είναι σημαντικά ποσά, να δαπανούνται με το καλύτερο τρόπο και να βοηθούν τις κοινωνίες αυτές να αναπτυχθούν σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχουν παγίδες και πολλές φορές όταν παίρνουμε το λόγο, όταν μιλάμε για απασχολησιμότητα, για ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε χιλιάδες πτυχία, διπλώματα και δεξιότητες σε τομείς οι οποίοι δεν υπάρχουν πια όταν οι άνθρωποι αυτοί φτάσουν στην αγορά εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την προσοχή σας και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την ακρόαση.